Τετάρτη 26 του μηνό. Αν δεν διαφωνεί κανένας, συμφωνούμε την εμμυρισία διάταξη. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, έχουμε τώρα τη μεγάλη τιμή να καλωσορίσουμε τον Υπουργό κ. Σάντορ Πίντερ, Υπουργό Εσωτερικών της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι σήμερα έχουμε δύο υπουργούς της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα αρχίσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατά νου το γεγονός αυτό για να αποφευχθούν κατά δυνατόν οι επικαλύψεις ή αναμίξεις ερωτήσεων που σχετίζονται με άλλους τομείς δράσης της Ουγγρικής κυβέρνησης όπως παραδείγματος χάρη δικαιοσύνη, κοινωνική ένταξη, μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένο και το θέμα της ένταξης των ΛΟΜΑ, θέμα που θα εξεταστεί με άλλο εκπρόσωπο της Ουγγρικής κυβέρνησης που θα καλωσορίσουμε προσεχώς εδώ σήμερα και τις επόμενες μέρες. Έχουμε δύο υπουργού σήμερα και έχουμε και κάποια άλλα θέματα στη ημερησία μας διάταξη, ίσως ίσονος σημασίας. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους χρονικούς περιορισμούς που έχουμε. Θα πρότεινα ο Υπουργός να κάνει την παρουσία του σε 10, το πολύ 15 λεπτά μετά θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συνονιστές, ο καθένας δύο λεπτά. Μετά θα απαντήσει ο υπουργό κ. Σάντορ Πίντερ. Και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ανοιχτό για όποιους βουλευτές θέλουν να πάρουν το λόγο. Και τελικά θα υπάρχει και χρόνο για τον Υπουργό. Έτσι, θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σε μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο, όχι περισσότερο γιατί έχουμε και άλλο υπουργό που θα έρθει και έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα. Έχουμε πάρα πολύ βεβαρημένη μέσα διάταξη σήμερα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και σας δίνω το λόγο. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlament! Nagyon örülök, hogy a magyar kormánynak Αγαπητά μέλη, χαίρομαι διότι έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις ε, προτεραιότητες εσωτερικής πολιτικής της Ουγγρικής Προεδρίας. Και χαίρομαι διότι θα έχω την ευκαιρία να σας πω πώς βλέπουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης θέτει τις βάσεις συνεργασίας. Και μέσα στα πλαίσια της θέσης σε εφαρμογή θα θέλαμε να εξετάσουμε όλες τις προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος η πρώτη μας προτεραιότητα. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συζητήθηκε από το Συμβούλιο το 2000 και θεωρήσαμε ότι έχει παρέλθει μία δεκαετία πλέον, οπότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το συζητήσουμε εκ νέου. Έχουμε πολλούς λόγους για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Ζήσαμε μία μεγάλη κρίση δεν έχουμε ανακάμψει πλήρως από αυτήν, η οποία έχει πλήξει όχι μόνο την οικονομία, τις αξίες μας, αλλά έχει επιπτώσεις και στο οργανωμένο έγκλημα. Συνεπώς θα πρέπει να αναλύσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στο οργανωμένο έγκλημα και να δούμε πώς θα ανταποκριθούν τα μεμονωμένα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση. Η εργασία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Βασιζόμαστε στη Europol, στη Frontex και στα κράτη-μέλη. Έχουμε καταρτήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο υποβάλαμε και συζητήσαμε σε επίπεδο Συμβουλίου. Το Συμβούλιο στο Συμβούλιο αυτό ο κύριος Λόπες Αγκουιλάρ έλαβε το λόγο και συνεισέφερε στη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Μίλησε για τακτικότερη και στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι πολύ σωστά επιλέξαμε αυτήν την προτεραιότητα. γιατί χρησιμοποίησαμε το πρόγραμμα της ε, Στοχόλμης ως βάση, καθώς και την ε, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας που εγκρίθηκε πέρσι το Μάρτιο καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής που εγκρίθηκε το Νοέμβριο. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ορισμένα σημεία κλειδιά. Ένα από αυτά είναι η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. Και θα ήθελα να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημασία η ροή πληροφοριών διότι ε, ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες όχι μόνο μέσω Europol. Υπάρχει ένα κέντρο συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με κέντρο το Βουκουρέστι και νομίζω ότι το ΣΕΦΙ θα διαδραματίσει πολύ ε, σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πιστεύω ότι το, οι πληροφορίες αυτού του κέντρου θα πρέπει να μεταβιβάζονται στη Europol. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση των Βαλκανίων στα Βαλκάνια και αυτό συνεισφέρει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η νέα προτεραιότητα, η επόμενη προτεραιότητα είναι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων διότι έτσι θα υποσκάψουμε τα θεμέλια του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν θα υπάρχουν ε, περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσει να δράσει το οργανωμένο έγκλημα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή χρηματοδότηση, επαρκής ε, χρηματοδότηση. Αυτές είναι οι οικονομικές βάσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης υπάρχει η σύσταση μια ομάδας με κράτη-μέλη, Europol και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντάξουμε ένα εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο θα ασχοληθεί με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε ότι όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα κατά συγκεκριμένους τρόπους. Υπάρχει όμως διαφορετική αντιμετώπιση από κράτος σε κράτος. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι βέλτιστες δυνατές πρακτικές και οι καλύτερες απαντήσεις για να δώσουμε απάντηση. Στη συνάντηση του Συμβουλίου ζήτησα τη συνεργασία όλων των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών και του ζήτησα να ε, διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα που θα ασχοληθεί με αυτό το εγχειρίδιο για να δούμε την εγκληματική συμπεριφορά και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Αυτό το εγχειρίδιο λοιπόν θα ασχοληθεί με την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στα επιμέρους κράτη-μέλη. Επίσης, μας ενδιαφέρει η, ανατολικές, η ανατολική οι ανατολικές εταιρικές σχέσεις. Δηλαδή κοιτάμε πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και ιδέες σε αυτούς τους τομείς. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι οι ανατολικοί μας εταίροι θα μπορέσουν να ασχοληθούν με θέματα παράνομης μετανάστευσης. Θα έχουμε δηλαδή ένα μηχανισμό φιλτραρίσματος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αποφορτίσουμε την κατάσταση από εμάς. Και να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας για να φτάσουμε σε ευρωπαϊκές ε, προδιαγραφές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι ύψιστης της σημασίας για μας είναι η Συμφωνία Σέγγεν και η προσχώρηση δύο χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Θα προσχωρήσουν στη Συμφωνία Σέγγεν όπως γνωρίζετε στο εγγύς μέλλον. Αυτό το θέμα το έχουμε θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων μας και όταν μας ε, πρώτα απασχόλησε, είδαμε ποια είναι τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων. Είδαμε ότι οι δύο αυτές χώρες πληρούν τους όρους και μπορούμε να έχουμε θετικά, θετική έκβαση. Πρόσφατα, στις πρόσφατες συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες γνωρίζουμε ότι η Βουλγαρία δεν πληρεί όλους τους όρους η Ρουμανία πληρεί τα, τις τεχνικές προδιαγραφές, γιατί μιλώ μόνο για τις τεχνικές προδιαγραφές επί του παρόντος. Γιατί στα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας δεν υπάρχουν έλεγχοι, άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύο χώρες ξεχωριστά. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε από τη Βουλγαρία μέχρι ότου πληρεί τους όρους για να μπορέσουν να ενταχθούν και οι δύο χώρες. Ο Υπουργός Εσωτερικών της ε, Βουλγαρίας εκπροσωπήθηκε και μας είπε ότι θα προσπαθήσει να συμμορφωθεί προς τους όρους μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε χώρες, οποιαδήποτε χώρα να προσχωρήσει αν δεν πληρεί τους ε, όρους 100%. Έλαβα δύο επιστολές από τους υπουργού εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας που αντιτάχθηκαν στην προσχώρηση των δύο αυτών χωρών στη Συμφωνία Σέγγεν διότι υπάρχει θέμα διαφθοράς δικαιοσύνης και ούτω καθεξής όπου δυστυχώς ε, τα εχέγγυα δεν είναι πολύ καλά από αυτές τις δύο χώρες. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που με απασχολούν, γι' αυτό θα ήθελα να επιταχύνω κάπως. Η συμφωνία PNR μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για τα στοιχεία δηλαδή επιβατών, για τα στοιχεία επιβατών, νομίζω ότι ακολουθούμε έναν πολύ καλό ρυθμό, αλλά μας ενδιαφέρει και η, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Αυτές είναι προτεραιότητες που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη δεν είναι θέμα αρμοδιότητας του Συμβουλίου, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο βασικός διαπραγματευτής. Θα πρέπει όμως να υποστηρίξουμε την Κομισιόν στις προσπάθειές της. Ένας άλλος σοβαρός ε, τομέας είναι να συσταθεί το σύστημα Eurodec. Σε σχέση με την νόμιμη μετανάστευση υπάρχουν αρκετά θέματα το θέμα της ενιαίας άδειας παραμονής είναι ένα από τα θέματα. Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά. Μετά μιλάμε για τα, τους εποχικούς εργαζόμενους και το, τις εποχικές άδειες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί. Και μιλάμε και για μετα, μεταφορές ICT, δηλαδή μεταφορές μεταξύ επιχειρήσεων. Εδώ βρισκόμαστε σε συμφωνία με το Συμβουλίο. Όλοι οι Υπουργοί Εσωτερικών συμφώνησαν και δέχτηκαν τα, την ύπαρξη των ICT των μεταφορών δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και το θέμα της ενιαίας άδειας παραμονής μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και σε αυτόν το τομέα. Ένα άλλο σημαντικό σύστημα είναι το VIS, το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων για τις θεωρήσεις. Υπάρχει προθεσμία του Ιουνίου, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή καθώς και το SIS-2, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, το δεύτερο πρόγραμμα, η, η Ουγγαρία ήταν υποψήφια χώρα όταν είχε πρωτοτέθει το ζήτημα. Το ΣΥΣ 2 τότε είχε ξεκινήσει. Ελπίζω να αποτελέσει πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στη στρατηγική του Δούναβη, διότι έχουμε πολλά να κάνουμε να επιτελέσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Ο Δούναβης είναι η έβδομη μεγαλύτερη πλωτή οδός. Θα θέλαμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών και επίσης να μην μεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επαυξημένη εποπτεία, να ασχοληθούμε και με τα θεμελιώδη δικαιώματα και βασιζόμαστε στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να εξορροπήσουμε τα δύο σκέλη. Εάν το καταφέρουμε αυτό, θα θεωρήσουμε ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχής προεδρία μας. 12,5 λεπτά μίλησα μόνο, άρα είμαστε στην ώρα μας για τις ε, ρωταποκρίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό για την παρουσίασή του αυτή. Ευχαριστούμε που σεβάστηκε και την πρόταση για τον περιορισμό του χρόνου. Θα κάνουμε τώρα ένα πρώτο γύρο των συντονιστών, όπως είπαμε. Εξονόμητος του ΕΛΚ τώρα. Ο Καλός θα πάρει το λόγο. Δύο λεπτά θα έλεγα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό, να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του και θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, λυπάμαι διότι δεν θα παρευρεθώ καθ' τη διάρκεια της συνεδρίασης. Γίνεται μια κρόαση και στην Υποεπίτροπη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις προς τον Υπουργό σε σχέση με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η ερώτηση ίσως φανεί ρητορικής φύσης, αλλά δεν είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι κατά την Προεδρία σας θα πρέπει να μπουν αυτές οι δύο χώρες στον ε, χώρο Σέγγεν είναι προτεραιότητα για σας και εάν ναι, πώς θα συνεργαστείτε έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις. Όπως είπατε στην παρουσίασή σας, θα θέλαμε να ενταχθούν οι δύο χώρες στο χώρο Σέγγεν, αλλά αυτό ε, αφορά ορισμένες προαπαιτήσεις ασφάλειας. Θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στις ε, εκθέσεις αξιολόγησης. Τις έχουμε ζητήσει ήδη. Δεν μας πάτησαν το Συμβούλιο επίσημα και άτυπα μάθαμε ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά μας, διότι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο πολύ λίγοι βουλευτές, δηλαδή μόνο οι σκιώδεις. οι Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για το Κοινοβούλιο. Το δεύτερο ερώτημα έχει σχέση με το ΣΥΣ2, το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο ΣΥΣ κατά την εξάμηνη προεδρία σας. Ως προς το ΕΡΟΝΤΑΚ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στον τομέα των βασικών ελευθεριών και δικαιοσύνης θα θέλαμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Πιστεύετε ότι κατά την εξάμηνη προεδρία σας θα σταθεί αυτό δυνατόν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Chairman, and thank you, Minister, for... Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την τόσο πλήρη αυτή παρουσίαση. Καλύψατε πάρα πολλούς ε, τομείς, ε, κύριε Υπουργέ. Δεν θα υποβάλω δύο ή μάλλον τρεις ερωτήσεις για ένα πιο ε, αμφιλεγόμενο και δύσκολο τμήμα Προεδρία σα. Στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια καλή και λεπτομερή συζήτηση για το θέμα του ασύλου. Και χαιρόμαστε που σε αυτό αφιέρωσε η Προεδρία ε, κατά την παρουσίασή σε ένα σημαντικό τμήμα του χρόνου που είχε. να να αναφερθώ στις διαδικασίες ε, που θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν όπως είπατε πλησιάζουμε την ε, προθεσμία του 2012 για τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασυλίας και βλέπουμε ότι τα κρατημέρια στο Συμβούλιο ανησυχούν για το κόστος Φερρυπίν. Είπαμε πολλές φορές ότι το θέμα της ποιότητα των αποφάσεων που θα ληφθούν, το λεγόμενο fraud logging και η διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά και είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση από την Προεδρία στην Αραμέλη την περασμένη εβδομάδα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για τις προτάσεις σας για το συνολικό, ε, τη συνολική αυτή δέσμη και για το Eurodoc. Δεύτερον, Αναφέρεται αρκετά λεπτομερό στο θέμα του οργανωμένου εγκλήματος και της στρατηγικής εσωτερικής στρατηγικής. Χαιρόμαστε που τονίζει το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, το θέμα κατά της ε, μαφίας ε, που ετέθηκε και ε, αυτή για το θέμα του Σέγγεν, δεν θέλω λοιπόν να επαναλάβω, για την Ευρωπόλ μόνο. Θα θέλαμε να υπάρξει πρόοδος και πραγματικέ αποφάσεις. Πολύ καλή λοιπόν αυτή η δήλωσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαράης των Σοσιαλιστών, η ομάδα Άλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Υπουργέ που μας παρουσιάσατε αρκετά μακρύ κατάλογο θεμάτων που αφορούν ε, και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε ότι αυτά είναι τμήματα των προτεραιοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω καλύτερα ποια είναι η θέση της Ουγγρικής Προεδρίας όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα. αναφέρθηκατε στην ιδέα της καταπολέμησης της παράνομης ε, μετανάστευσης εκτός των συνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν περόδο αναφερθήκατε και στην ιδέα ε, της ε, νόμιμης μετανάστευσης επίσης. Θα ήθελα να ξέρω η Ουγγρική Προεδρία έχει προτεραιότητα ε, <clears throat> έγκρισης του φακέλου αυτού για την ενιαία άδεια για τους ε, εποχιακά εργαζόμενους που θα ισχύει για όλη την Ένωση. Επίσης, ποια είναι η θέση της Ουγγρικής Προεδρίας όσον αφορά την πρόσβαση των ε, υπηρεσιών καταστολής εγκλήματος στα στοιχεία του Eurodoc. Σέγγεν και η ένταξη των δύο εν λόγω χωρών στο χώρο Σέγγεν αναφέρατε ότι λάβατε δύο επιστολές από δύο υπουργούς που ήταν κατά αυτού. Αλλά θα ήθελα να ξέρω η δική σας, η ουγγρική θέση για το θέμα ποια είναι για τις δύο αυτές επιστολές. Και πάντα για το Σέγγεν θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε και ο κύριος Κοέλιο. Κατά τη γνώμη μας είναι απολύτως απαράδεκτο να μην επιτρέπεται στο Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε έγγραφα όταν εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Έτσι μας συμπεριφέρεται το Συμβούλιο. Και θα πρέπει νομίζω όμως να τύχουμε συμπεριφορά σε επίσης ώρες. Ευχαριστώ. Ξενόματος τον Πρασίνο κύριο Σαργεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να περάσω αμέσως στο θέμα ασύλου και μετανάστευσης είχατε την πρώτη ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την περασμένη εβδομάδα στην ε, Ουγγαρία και εκτός αυτού ε, λήφθη αυτή η απόφαση την περασμένη εβδομάδα για τους κρατούμενους βάση με το Δουβλίνο και ότι αυτή τη στιγμή δεν θα επιστρέφονται πια ε, στην Ελλάδα τα άτομα αυτά μου φαίνεται ότι είναι καλή απόφαση, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ε, μεγα, πολύ έντονος επίγον χαρακτήρας όσον αφορά τα θέματα της λειτουργίας της συνθήκης του Δουβλίνου. Την περασμένη εβδομάδα τι είπανε οι υπουργοί για το θέμα αυτό, γιατί αν κοιτάξω και τα δικά σας σχέδια για το, το, το εξάμεινο και την ημερησία διάταξη το χρονοδιάγραμμα μάλλον των συναντήσεων του Συμβουλίου, βλέπω ότι η επόμενη συνάντηση που έχετε είναι για τον Ιούνιο και για το άσυλο και τη μετανάστευση αναφέρεται state of play. Πού βρίσκονται τα πράγματα. Πού βρίσκονται λοιπόν τα πράγματα και πού θα ληφθούν και πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις. Το ότι δεν πρόκειται να επανασταλούν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη νομίζω να βρουν μια λύση για το Δουβλίνο. Και αναρωτιέμαι κατά πόσον και εσείς όπως και οι προηγούμενες προεδρίες έχετε έναν κατάλογο οδηγιών που πιστεύω ότι θα μπορείτε να προωθήσετε το επόμενο εξάμεινο. Κατόπιν και ακολουθώντας τις παρατηρήσεις κυρίας Βέμπερ, θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα ακόμα όσον αφορά τις την ε, σχέση της ανατολικής, ε, με τις ανατολικές χώρες και τον μηχανισμό φιλταρίσματος όπως κατάλαβα για την παράνομη μετανάστευση. Τι εννοείται με αυτό. Ευχαριστώ. Ξέρω μας CCR. Υπάρχει κάποιος εδώ που θα θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ταφάρης. ξέρω με Γκουε. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα υποβάλω τις ερωτήσεις μου στα πορτογαλικά. Μιλήσατε για θέματα παράνομης μετανάστευσης επί μακρόν. Αλλά απογοητεύτηκα κάπως διότι δεν έγινε ευρεία μνήα στα θύματα της παράνομης μετανάστευσης και πώς το Συμβούλιο υπό την Ουγγρική Προεδρία θεωρεί ότι θα μπορέσει να προστατεύσει τα θύματα της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας προσώπων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δίκτυα αυτά βασίζονται στους πρόσφυγες τι θα γίνει ως προς την ε, επανεγκατάσταση, resettlement και την απάντηση που αναμένουμε από το Συμβούλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι πολλές φορές αυτοί οι πρόσφυγες διέτρεχαν μεγάλους κινδύνους ως προς τη ζωή τους. Γι' αυτό έφυγαν από τη χώρα τους. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να επανεγκατασταθούν με τόσο μεγάλους κινδύνους. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το, την έκθεση την κοινή έκθεση με βάση την ε, διαδικασία συναπόφασης μέσα στα πλαίσια του ευρύτατου πολιτικού ε, φάσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή υπήρξε μεγάλη συμφωνία. Αναμένουμε μία απάντηση από το Συμβούλιο που δεν λάβαμε υπό Βελγική Προεδρία. Τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα πλέον ευάλωτα θύματα και θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσο η χώρα σας, ε, η Ουγγαρία, θα δράσει έτσι έστω και συμβολικά διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση τους Ουγγαρίας οδήγησε στη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Πώς θα αντιδράσετε σε αυτό το θέμα των θυμάτων? E για την EFD, κανένας, ναι, όχι, ωραία. Θα δώσουμε το λόγο για τους μία την κυρία Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύνηθες ότι όταν υπάρχει κάτι, ε, μια επίγουσα υπόθεση, μπορούν οι αστυνομικές δυνάμεις να περάσουν από τη μια χώρα στην άλλη. Εξωφρενικό μου φαίνεται αυτό. Είναι δεδομένο όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την νομοθεσία. Και σας ρωτάω τώρα, είναι δυνατόν σε μια παραδοσιακή δημοκρατία όπως στην Γαλλία ή στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιηθούν Ούγγροι αστυνομικοί όπως εκείνοι που επιτέθηκαν κατά ε, διαδηλωτών που επετέθηκαν στους στρατιωτικούς αυτούς και τους τραυμάτισαν άσχημα. Αθώους. Αυτή η αστυνομία που ξεπήρισε την δικτατορία που ήταν ε, επικεφαλής της χώρας για 8 χρόνια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Έχουν αποδιωχθεί τα άτομα αυτά από την ε, Ουγγρική αστυνομία και αν όχι γιατί όχι. Δεύτερον, πώς βλέπετε εσείς τις δράσεις κατά της τρομοκρατίας. Πώς σχετίζονται αυτά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο. Στην Ουγγαρία πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα νέο νομοσχέδιο που συμπεριλαμβάνει τον όρο άτομο σχετικό με την τρομοκρατία. που μπορεί να διωχθεί χωρίς δικαστική απόφαση. Εγώ, ως Ευρωβουλευτής, μπορώ να είμαι αντικείμενο τέτοια συμπεριφοράς, τέτοιων επιθέσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ολοκληρώσαμε το πρώτο γύρο για τις αντιδράσεις για τον Υπουργό και θα περάσουμε μετά τις απαντήσεις στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Köszönöm szépen, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις τους. Καταρχάς, κύριε Κοέλιο, το ερώτημά σας ήταν ποια είναι η θέση, η πραγματική θέση της ε, Ουγγαρίας για την ε, ένταξη στην, ε, χώρο Σέγγεν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Εμείς υποστηρίζουμε την ένταξη αυτών των δύο χωρών στον χώρο Σέγγεν. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι θέλουμε αυτές οι δύο χώρες να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια. Μόνο τότε θα μπορούν να ενταχθούν στο Σέγγεν. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρηθούν. Ο κανόνας λοιπόν λέει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να πληρεί όλα τα τεχνικά κριτήρια και μετά μπορεί να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Αυτή είναι η θέση μας και νομίζω ότι είναι αρκετά σαφής. Είναι σαφές ότι με βάση και τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων η... στα, στα, σύνορα... Στα... στα σύνορα με την Τουρκία, μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Και αυτό βέβαια δεν το λένε μόνο οι εμπειρογνώμονες αλλά και άλλοι. και άλλοι αξιωματούχοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, ακόμη και ο ίδιο ο Υπουργό Εσωτερικών το έχει παραδεχθεί. Και όπω είπα, υποσχέθηκαν ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα λύσουν το πρόβλημα και θα πληρούνται έτσι όλα τα κριτήρια για να μπορέσουν να ενταχθούν. Οπότε, αυτή τη στιγμή γίνει αυτό, μπορούμε να κάνουμε άλλη μία ανάλυση, να κάνουν άλλη μία ανάλυση οι για να δουν αν όντω πληρούνται τα ε, κριτήρια αν συμβαίνει αυτό, τότε εμεί θα υποστηρίξουμε την ένταξη των δύο χωρών. Επίση, η πρόσβαση των μελών του Κοινοβουλίου στι πληροφορίε των συμβουλίων, σε έγγραφα εμπιστευτικά, σε άλλε τέτοιε πληροφορίε, Έχω λάβει κάποια ενημέρωση ω προ αυτό, η οποία λέει ότι εάν είσαστε στο Συμβούλιο, έχετε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, αλλά το Συμβούλιο δεν μπορεί να στείλει τα έγγραφα αυτά στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Προσπαθώ να βελτιώσω με κάποιο τρόπο την κατάσταση για το μέλλον και θα ήθελα όντως αυτά τα έγγραφα στο μέλλον να παρέχονται στο Κοινοβούλιο τηρώντας βέβαια πάντα τις διάφορες δεκλίδες ασφαλείας που υπάρχουν και τα κριτήρια και την εμπιστευτικότητα κτλ. Να μπορούν όμως σε κάποια άτομα αυτά τα έγγραφα να αποστέλλονται, ειδικά σε ευρωβουλευτές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να έχουν τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα. Ε, πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει από το 2013. Το Συμβούλιο συμφωνεί, οι Υπουργοί Εσωτερικών συμφωνούν ότι αυτό το σημείο θα πρέπει να μείνει στις ημερήσεις διατάξεις, ακόμη και άτυπα, αλλά κάθε φορά θα πρέπει σε κάθε Συμβούλιο να ελέγχεται η πρόοδος που έχει γίνει, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε την πίεση. Αυτό εννοούσα ότι πρέπει να υπάρχει μια χρονικά δόκιμη εφαρμογή του συστήματος για την προστασία δεδομένων. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Όλες οι απαιτήσει προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να πληρούνται. Κανένα σύστημα δεν θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί εάν δεν πληρούνται όλες οι ε, απαιτήσει και τεχνικές και προσωπικές. Οπότε προφανώ πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια αυτά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να τέθει σε λειτουργία ένα σύστημα. Ο κύριο Μόρε έθεσε κάποια ερωτήματα. Νομίζω ότι αναφερθήκατε και στο πακέτο για το άσυλο. και είπατε ότι υπάρχει έτσι μια ανησυχία για το κόστος. Προφανώς όλοι επηρεαζόμαστε για το θέμα, από το θέμα αυτό. Ε, στο τελευταίο συμβούλιο, ε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, καθώ επίση και η ανάλυση που γίνεται για τα υπάρχοντα ε, χρηματοδοτικά μέσα και επίση συζητήσαμε το ποιε είναι οι προτεραιότητε και ποια είναι τα διαθέσιμα κονδύλια που έχουμε για να τα διαθέσουμε με σωστό τρόπο. Η Eurodac τώρα και η πρόσβαση στο σύστημα αυτό. Θα έλεγα ότι η αντιμετώπιση της, ε, του οργανωμένου εγκλήματος είναι μία από τις ε, πρώτες μας προτεραιότητες, ε, οι ποινικέ διώξεις, από την πλευρά μάλλον της ποινική δίωξης, οι διοκτικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα συστήματα αυτά, αλλά Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να καταστατηγήσουμε τελείως την ιδιωτικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά αν υπάρχουν ε, πληροφορίες για άτομα που, έχουν, ε, που κάνουν εμπόριο ε, ανθρώπων ή μπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, τότε προφανώς θα πρέπει οι διεκτικές αρχές να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω στις 10 Αυγούστου ήταν, αν θυμάμαι καλά, ε, Μάλλον στις 10 Αυγούστου θα είναι η μέρα που θα ε, τεθεί σε εφαρμογή η σύμβαση που έχει υπογραφεί ε, για την πρόσβαση σε λεπτομέρειες όπως ε, DNA, ε, δαχτυλικά αποτυπώματα, άλλα δεδομένα Αυτά είναι τα βασικά σημεία τη ε, σύμβαση αυτή. Η Ουγγαρία μπορεί να πλήρει τι προποθέσει που απαιτούνται μέχρι τι 10 του Αυγούστου. Θα είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Η βάση δεδομένων για το DNA είναι έτοιμη. Η βάση δεδομένων για τα συγκεκριμένα δεδομένα των ατόμων είναι έτοιμη. Για τα αποτυπώματα τώρα ε, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση τη ε, βάση δεδομένων μα. Οπότε μέχρι τον Αύγουστο θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε νομίζω ή ελπίζω τα περισσότερα κρατημέλη να μπορούν να το πράξουν, να πράξουν κάτι ανάλογο. Υπάρχουν όμω τέσσερα κράτη-μέλη, τα οποία ήδη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα. Ε, φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10 Αυγούστου θα υπάρξουν και άλλοι που θα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα κρατημέλη, λόγω οικονομικών δημοσιονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα κρατημέλη, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν σε αυτή τη σύμβαση και να μπορέσει η σύμβαση να τεθεί σε εφαρμογή. Το επόμενο ερώτημα για την νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Για την μετανάστευση Αυτό έχει γίνει, η λαθρομετανάστευση έχει γίνει η γραμμή παραγωγής του οργανωμένου εγκλήματος. Απαντώ και σε ένα άλλο ερώτημα έτσι, ε, που νομίζω το έθεσε ο κύριος Τάβαρες ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από χώρες που, ε, που κινδυνεύουν. Νομίζω ότι αυτές, οι, αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν όπου και αν είναι. Και πραγματικά κινδυνεύουν πάρα πολλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Στον ε, ποταμό Τίσα, ε, πολλές φορές στην Ουγγαρία, έχουμε δει ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν τον ποταμό με βάρκες, να πνίγονται στο ποτάμι, ούτως ή άλλως και, και εκεί που ήταν κινδύνευαν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για να φύγουν από εκεί πάλι κινδυνεύουν. Ένας άνθρωπος έχει επιβιώσει από αυτή την προσπάθεια ε, πλεύσης του ποταμού. Νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται μόνο για οικονομικούς λόγους στις ε, χώρες μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ούτως ή άλλως πρέπει να λάβουν βοήθεια. Ε, εμείς ε, Έχουμε υπόψη μας το θέμα αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε και άτεγκτοι εναντίον αυτών των ε, ε, εμπόρων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά εκμεταλλεύονται ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν ούτε καν τα χρειώδη και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στις ποινές που τους επιβάλλουμε, γιατί ουσιαστικά είναι έμποροι ανθρώπων. Τώρα, για την ενιαία άδεια. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Οι εποχιακοί τώρα ε, εργαζόμενοι και η σχετική άδεια υπάρχουν πολλά κρατημέλη που την υποστηρίζουν και εμείς την υποστηρίζουμε παρόλο που θεωρούμε ότι δεν είναι όσο αποτελεσματική είναι άλλες άδειε. Και το δύσκολο ερώτημα πόσο κρατάνε αυτές οι εποχές κατά τις οποίες εργάζονται οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Δηλαδή μιλούμε για τη συλλογή φρούτων για λίγες εβδομάδες, μιλούμε για, αν μιλούμε για άλλες, ε, ε, για άλλες ε, ας πούμε για τις, για τις κατασκευές μπορεί το έργο να κρατήσει και ένα χρόνο και δύο και αυτό να θεωρείται πάλι εποχιακή εργασία. Οπότε πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά γιατί οι προποθέσει αυτές θα πρέπει να θα επηρεάσουν και, τους, και τις οικογένειες των εργαζόμενων αυτών. Εκεί έγκυται οι περισσότερες ε, διαφορές που υπάρχουν στις απόψεις στο Συμβούλιο. Αυτά τα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα σε ένα πακέτο ούτε από το Κοινοβούλιο νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν να τα δούμε ξεχωριστά ένα προς ένα, γιατί συμφωνούμε για τις ε, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και τα ICTs. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο εάν μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Και έχουμε και άλλα δύο θέματα, την, ε, τους επιχειρικούς εργαζόμενους και την ενιαία άδεια. Εάν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το ένα από τα τρία αυτά θέματα, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Αν ας πούμε μπορέσουμε να δούμε το θέμα τη ε, ενία άδειας, θα μπορέσουμε προφανώ να λύσουμε και κάποιε πτυχέ του θέματο των εποχιακών εργαζομένων. Τώρα, για την προστασία, για την πρόσβαση στα δεδομένα από τι δικτικές αρχέ. Δεν νομίζω ότι το φιλτράρισμα των δεδομένων είναι καλή ιδέα. Αλλά Εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση, μια συγκεκριμένη υπόθεση, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Ούτε οι ίδιε οι ιδιοκτικέ αρχέ θα πρέπει να εθελοτυφλούν. Θα πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλε αυτέ τι πληροφορίε και τα δεδομένα. Αυτέ οι ε, αρχέ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και όχι γιατί είναι περίεργες αλλά είναι, είναι ε, αρμοδιότητά του να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Εσάς τα παιδιά σας να κάνουν την ζωή σας πιο ασφαλή. Αυτή είναι η, η δουλειά των αρχών επιβολής του νόμου και νομίζω ότι θα πρέπει να τους δώσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουν για να το πράξουν αυτό. Πάμε πάλι πίσω στη Σέγγεν. Να τονίσω και πάλι ότι εμείς υποστηρίζουμε την πρόσβαση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν, αλλά περιμένουμε και από τις δύο χώρες να ανταποκριθούν στις τεχνικές ε, προδιαγραφές που υπάρχουν και τις οποίες πληρώνουν όλα τα υπόλοιπα κρατημέλη. Η κυρία Σαργεντίνη ρώτησε για το δικαστήριο και για τον κανονισμό Δουβλίνο. Ε, θα είμαι... τι θέλετε να σταματήσω, πρόεδρε? Α, ωραία. Ναι, θα είμαι σύντομος. Ε, μου έδωσε ο πρόεδρος λίγο χρόνο ακόμη. Λοιπόν, Δουβλίνο. και σε ό,τι αφορά το θέμα της Ελλάδας. Υπάρχουν 40.000 παράνομοι μετανάστες, τους οποίους δεν μπορεί να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος. Εμείς τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε πάρει ένα προσωρινό μέτρο. Στείλαμε στρατιωτικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και Ούγγρους, για να υποστηρίξουν την, ε, τις ε, ελληνικές αρχές. Ε, μειώθηκε λοιπόν κατά 40% η ελευθερομετανάστευση μετά από την αποστολή αυτών των μονάδων, οπότε αυτό είχε ε, αποτέλεσμα. Το δικαστήριο στο Στρασβούργο μα έδωσε κάποια καθοδήγηση. Τώρα ε, θα τηρήσουμε όλε τι αποφάσει του, του δικαστηρίου, θα αναθεωρήσουμε την κατάσταση όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα, σχέσει με ανατολικέ με ανατολικές χώρες, υπάρχουν έξι χώρε στα, σύνορα ε, στα ανατολικά σύνορα της, Ευρώπη, ε, Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία Γεωργία, Αρμενία, όλες αυτές οι χώρες έχουν τα ίδια προβλήματα. Εάν ε, χρησιμοποιούσαν την, ε, την ίδια ε, προσέγγιση απέναντι στην λαθρομετανάστευση, στο εμπόριο ανθρώπων κτλ. θα μπορούσαν ίσως να σταματήσουν αυτές τις ροές και να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες αρχές όταν αξιολογούν την κατάσταση όπως κάνουν και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Αυτό θεωρώ εγώ ως φίλτρο, γιατί αυτές οι ροές σταματούν και ταυτόχρονα συμβάλλουμε και στην ενίσχυση του νομικού συστήματος, του συστήματος δικαίου αυτών των χωρών, γιατί έτσι θα ε, προσεγγίσει λίγο τα συστήματα δικαίου των δικών μας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1956 Ο υπότος αρμοστής για τους πρόσφυγες στον ΟΗΕ είχε μια έδρα στο, είχε γραφείο στο, στην Ουγγαρία και είχαμε λάβει ε, πολύ καλή καθοδήγηση τότε για το θέμα αυτό από, το, από τον ίδιο. Τώρα για τις αστυνομικές δυνάμεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, το έχετε δει αυτό και στην ε, Ουγγαρία. Έχετε δει πολλούς, πολλές αστυνομικές δυνάμεις ε, να κινούνται σε διάφορες πόλεις όταν υπάρχουν μεγάλες ε, ροές τουριστών και υπάρχουν και άλλοι, άλλες μονάδες από άλλες χώρες που έρχονται να βοηθήσουν ε, και βοηθούν τους τουρίστες. Αλλά και οι Ούγγροι αστυνομικοί που πάνε πολλές φορές στην Κροατία για να βοηθήσουν τους Ούγγρους τουρίστες στην Κροατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Εγώ έχω πάει στην Βαβαρία και είπαμε ότι κατά τη διάρκεια του Oktoberfest θα πηγαίνουν αστυνομικοί Ούγγροι για να βοηθούν τους τουρίστες από την Ουγγαρία εκεί ώστε να μην, να μην φοβούνται, να μην νιώθουν ασφάλεια. Και νομίζω ότι στην Ουγγαρία σε σύγκριση ε, μέσα στο, στην 8 ετία 2002-2010 τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Έχουμε αλλάξει την ιδεολογία, την οτροπία των αστυνομικών δυνάμεων και όσοι δεν συμφωνούσαν στην, ε, ε, με την αλλαγή αυτή, στην ιδεολογία και στην ε, προσέγγιση, έφυγαν από το σώμα. Οπότε νομίζω ότι προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αντιμετώπιση τρομοκρατίας και ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Οι χώρε που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία, πολλές φορές κινούνται προς το να ε, στοχεύσουν μόνο σε αυτό, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και παραβλέπουν λίγο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Αντιμετώπιση εγκλήματος, αντιμετώπιση τρομοκρατίας, απ' την άλλη όμως προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Ένα λεπτό, κύριε Ταβάλα. Στι 10 ε, έχουμε τον Υπουργό Ζόλταν Πάλοκ που θα εξετάσει το θέμα της κοινωνικής ένεξης και των Ρωμά. Λοιπόν, θα έλεγα... Θα σας διαβάσω εδώ τον, να κάνουμε το δεύτερο γύρο, έχω τον κατάλογο, παρακαλώ. Díaz de Mera, Hankis, Romero Lopez, Strasser, Interveld and McAvey. So I suggest that this second round is going to be one. Θα έλεγα λοιπόν ένα λεπτό καθένα στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει και ο Υπουργό να απαντήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ βεβαρημένη σε διάταξη ως συνήθω σήμερα. Το δικαστικό κύριε Ταβάρε. Ναι. Να διευκρινιστεί δεν ξέρω, ίσως δεν με καταλάβατε ή δεν καταλαβαινω τον Υπουργό. Εγώ ρώτησα κατά πόσον το ε, Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την διαδικασία συναπόφασης για την επανεκατάσταση. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, ελπίζω. Ελπίζω ότι θα γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο σύντομος. Λοιπόν, ένα λεπτό. Δεύτερο γύρο. Κύριε Σόλβερ, σας ευχαριστώ. Όπως και την περασμένη φορά, θα σας ζητήσω περισσότερο χρόνο. Γιατί μια που δεν είναι εδώ ο κύριος Μπουσουτήλ, με παραγκάλεσε να υποβάλω τις ερωτάσεις του ΕΛΚ για το σένκε καταρχήν. Τεχνικά κριτήρια υπάρχουν ε, με προβλήματα, αλλά υπάρχουν και τα πολιτικά κριτήρια. Ζητούμε λοιπόν καταρχήν να τεθούν τα σαφή κριτήρια γιατί η διαφορά, διαφθορά θα είναι ένα εμπόδιο της συνεργασίας κλπ. Αυτά για το Σέγγεν. Και θα συνεχίσω στα Ουγγρικά. Ασφάλεια και βασικά δικαιώματα. Θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένο η Frontex να μπορεί να εξετάζει τα προσωπικά στοιχεία. Ευρωπαϊκή Ελληνική. είναι σημαντικό να υπάρχουν δυνάμεις πρώτης κρούσεως στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναβληθούν περαιτέρω δράσεις. Το θέμα της ασυλία, του ασυλίου μπορεί να συμφωνήσει για οικονομική ενίσχυση το Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αλληλεγγύη που θα πρέπει να επιδείξουμε στα χτεσινά θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Θα ήθελα να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία. Προτεραιότητα είναι να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένα διασυνοριακό θέμα να καταπολεμήσουμε την δουλεία, το, την παραχάραξη του ευρώ, την παραχάραξη έργων τέχνης, ε, διακίνηση ναρκωτικών όλα αυτά αφορούν ένα ε, πλαίσιο πέρα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Europol δεν έχει κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει υπερεθνικό χαρακτήρα. Εσείς ως Ουγγρική Προεδρία θα προωθήσετε το νέο κανονισμό της Europol που θα δώσει νέες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα προωθήσετε τη διαδικασία αξιολόγησης της Europol έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα μέχρι το 2012 και μέχρι το 2013 να έχουμε τον νέο κανονισμό της Europol χωρίς νέες καθυστερήσεις. Κυρία Χάνκης. Ευχαριστώ. σε σχέση με την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, ως προς τις προτεραιότητες υπάρχει μια στρατηγική και ένα πρόγραμμα δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναθεωρείται κάθε χρόνο. Ε, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν και που είναι επιτάπητος, που τέθηκαν επιτάπητος πρόσφατα. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πέρα από το SWIFT και το PNR, τις πληροφορίες για, τις, για τους επιβάτες. Μέσα στα πλαίσια μη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που χρησιμοποιούνται ως προκάλημα για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα, πώς ε, αλληλοσχετίζονται. Υπάρχουν στοιχεία ότι οι τρομοκρατικές ε, ομάδες ε, ενδυναμώνονται από το οργανωμένο έγκλημα το ένα σκέλος ε, δρά με βάση η ιδεολογία, ενώ το άλλο με βάση τα κέρδη. Αλλά υπάρχει ένα είδος συνέργειας. Ως προς την ροή πληροφοριών, πώς μπορεί να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προωθήσετε αυτή την συνεργασία. Y κυρία Ρουμέρο επιμένω στο θέμα του πακέτου του ασύλου. Διότι συγχαίουμε τους παράνους μετανάστες και τους ετούντες άσυλο. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά ζητήματα. Γιατί όπως ξέρετε αυτοί που ζητούν άσυλο έχουν ε, ε, επιπρόσθετη κάλυψη. Ο ο ετών στο δικαστήριο του Στρασβούργου ζήτησε άσυλο με βάση τα δεδομένα της βελικής και της ελληνικής νομοθεσίας. Έγινε λόγος για 40.000 στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει και μία επικουρική κάλυψη, δηλαδή είτε θα διαγράψετε τον κανονισμό του Δουβλίνου, είτε θα δείτε ένα νέο, άλλο πλαίσιο αντιμετώπιση. Στράσε. Σας χαιρετώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε πολύ αναλυτικό πρόγραμμα στην Προεδρία σας που το παρουσιάσατε και μας ενδιαφέρει το θέμα ε, του ασύλου, της συμφωνίας BNR για τα στοιχεία των οξυδατών η στάση για το Schengen είναι κάτι που συμμεριζόμαστε σε μεγάλο ποσοστό έχουμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουν οι χώρες μέλη αλλά θα πρέπει να τηρούν και τα κριτήρια που έχουν τεθεί είναι ευχάριστο που ζητάτε καλύτερη συνεργασία του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο αυτό και ευκταίο και ως Αυστριακός εγώ χαίρομαι για τις δραστηριότητε για την ε, στρατηγική του, για το Δούναβι. Θα με διέφερε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπετε όσον αφορά την ασφάλεια, τον τέταρτο πυλώνα. Thank you. Mrs. Ευχαριστώ κύριε Ιντφέλντ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ γλίγορα. Τρεις ερωτήσεις το Συμβούλιο εθέτησε μία εντολή για να διαπραγματευτεί με τη ΣΥΠΑ για την ε, προστασία των ε, δεδομένων των διαταλλαγές ε, μεταφορές. Δεν έχει οριστεί όμως ο κύριος διαπραγματευτής θα επιταχύνει διαδικασία η Ουγγρική Προεδρία κατόπιν το θέμα της Eurodoc Αναφερθήκατε πολύ γρήγορα στο συσχετισμό μεταξύ τη ε, πολιτική ασούλου και οργανωμένου εγκλήματος. Σε μία πρόταση τα αναφέρετε και τα δύο. Γιατί, μήπω μπορείτε να μου πείτε. Και μια που δεν ξέρω ποιο είναι ο υπεύθυνο υπουργό, θα σα πω ότι στι 19 Φεβρουαρίου η Ουγγρική Προεδρία θα οργανώσει μια διάσκεψη για την οικογένεια και τα ποσοστά γενικότητα, αν κατάλαβα καλά. Τα κράτη-μέλη επιμένουν στην επικουρικότητα και γιατί θεωρούν ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σχέση με την οικογενειακή πολιτική και τα ποσοστά γενικότητα. Αν θεωρείτε ότι έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλαμβάνεται κάθου είδους ε, ε, οικογένεια. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. My question follows up. Η ερώτησή μου ακολουθεί το επόμενο ερώτημα για την καταπολέμηση του εργονομένου εγκλήματος και της νομοκρατίας και σχετίστηκε με διαφθορά γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία χωρίς διαφορά. Η Κομισιόν προσπαθεί να ολοκληρώσει μία ανακοίνωση για την κοινοτική πολιτική κατά της διαφθοράς. Και θα ρωτώ, θα υποστηρίξετε τις εργασίες της Κομισιόν σχετικά με την κοινωτική πολιτική κατά της διαφθοράς. Σκοπεύετε να υποστηρίξετε και να ενδυναμώσετε τις πολιτικές αυτές και ίσως να επιταχύνετε τη διαδικασία για την προετοιμασία της ανακοίνωσης. Πρώτα σας ευχαριστώ. Υπουργός έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο στις απαντήσεις μου. Καταρχήν, ως προς το πρώτο ερώτημα που σχετίζεται με το Σέγγεν, την ε, προσχώρηση στο Σέγγεν, το ερώτημα του κυρίου Σόγκορ. Είναι σαφές για μένα ότι έχουμε αναλάβει σαφή δέσμευση ως προς την προσχώρηση στο Σέγγεν. Μας απασχολεί βεβαίως και ο τομέας της ε, δικαιοσύνης και η επιστολή των Υπουργών Εσωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα υπάρχουν, αλλά ε, πρέπει να υπάρξει ομοφωνία από τα κράτη-μέλη για προσχώρηση στο Σέγγεν ως προς την αντιμετώπιση του Frontex στα ελληνικά σύνορα είχαμε μεγάλη επιτυχία. Μιλήσαμε για μείωση 40% σε σχέση με, τις, με την παράνομη είσοδο μέσω ελληνικών συνόρων μέσα στα πλαίσια ενός μήνα. Βεβαίως αυτό δεν είναι μια βιώσιμη λύση. Θα πρέπει να εξεύρουμε μια διαφορετική, ένα διαφορετικό σχήμα και ως προς την χρηματοδοτική αλληλεγγύη το διαπραγματευόμαστε, αλλά είναι πολύ δύσκολο την ε, παρούσα στιγμή να γίνει σωστή κατανομή κονδυλίων. Δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα πρότασης λύσεων στο Συμβούλιο. Το επόμενο, ως προς το επόμενο ερώτημα. Χτες το βράδυ στη Μόσχα έγινε μια τρομοκρατική ενέργεια, σκοτώθηκαν 30 και ε, είχαμε 135 τραυματίες από την τρομοκρατική αυτή ενέργεια. Θα ήθελα να εκφράσω τη, τη λύπη μου. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ενέργεια κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως προς την ε, Επιτάχυνση της διαδικασίας του νέου κανονισμού της Europol προωθώ όλες τις ε, δραστηριότητες προώθησης της ασφάλειας και η επιτάχυση της διαδικασίας Europol θα βοηθήσει στην ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Χάνκης μίλησε για το πρόγραμμα δράσης Υπάρχει ένα θέμα χρηματοδότησης για την στρατηγική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συζητήσαμε αυτό το θέμα γιατί κάτω από το 1% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δαπανάται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα ασφάλειας και να δούμε κατά πόσο τα κονδύλια αρκούν. Τώρα, ως προς τον συσχετισμό τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Η τρομοκρατία έχει μία ιδεολογική βάση, αλλά για να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους ε, χρειάζονται χρηματοδότηση, χρηματικούς πόρους, οι οποίοι πόροι δεν έχουν ιδεολογική βάση. Ε, βρίσκονται μέσω πώληση ναρκωτικών, εμπορίου όπλων και ούτω έτσι αγοράζουν όπλα οι τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Γι' αυτό υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας, διότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ παραγωγών ναρκωτικών, καλλιεργητών ναρκωτικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Η ιδεολογία είναι η τάση, αλλά το οργανωμένο έγκλημα προβάλλει τα μέσα. Έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο πάταξης της τρομοκρατίας στη Δυτική Ευρώπη και υπάρχουν ε, διάφοροι οργανισμοί στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το κέντρο θα ενταχθεί σε ένα δίκτυο παρομοίων κέντρων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ρομέρο ε, ρώτησε για το πακέτο αράνομη μετανάστευση. Είπε ότι αυτά τα δύο θέματα διαχωρίζονται. Όχι όμως απόλυτα. Εάν κάποιος έχει επανέλθει αρκετές φορές ως παράνομος μετανάστης, την τέταρτη πέμπτη φορά θα ετηθεί ασύλου. Αυτά τα θέματα λοιπόν αλληλοσχετίζονται. Υπάρχει συσχετισμός. υπάρχουν ε, ε, ετούντες ε, άσυλο του κλασικού τύπου, κλασικού τύπου που θέλουν να ξεφύγουν από μια επικίνδυνη κατάσταση στη χώρα προέλευσης τους και υπάρχουν βεβαίως και τυχοδιώκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα χορήγησης ασύλου και το καταχρώνται. Αυτό το θέμα θα το διαπραγματευτούμε και κατά την ε, Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και το θέμα της επικουρικής προστασίας και ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται σε αυτή την περίπτωση. Αυτό θα συζητηθεί και μέσα στα πλαίσια του Eurodac και του κανονισμού του Δουβλίνου. Θα θέλαμε αυτό το πακέτο να ε, φτάσει στη σέσιο πέρας ε, κατά την Προεδρία μας. Ο κύριος Στράσερ υπέβαλε ένα πολύ σωστό ερώτημα. Θα πρέπει να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές βεβαίως για την προσχώρηση στο Σέγγεν. Τώρα, ως προς τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, αυτό είναι ένα θέμα προτεραιότητας κατά την Προεδρία μας. Εάν ε, βλέπουμε τις ε, δικές μας χώρες, τη δική μας χώρα, χωρίς να ληφθεί μια απόφαση από το Κοινοβούλιο, τότε κανένας δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει οποιαδήποτε ε, δράση. Ως προς την στρατηγική του Δούναβη, αυτό είναι ένα θέμα προτεραιότητας. Εμείς έχουμε προβεί στη σύσταση ενός διαφορετικού οργανισμού με μια ξεχωριστή γραμματεία, αυτόνομη γραμματεία, για να λάβουμε υπόψη τις υποδείξεις ένταξη σε αυτή την πολιτική και με τη Σερβία και άλλες χώρες, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος να καλύπτει τον τομέα της ε, προστασίας και ασφάλειας σε αυτή την περιοχή, δηλαδή νότια του Δουνάβεως. Ως προς το PNR, της ε, διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ναι, υπάρχει η εντολή, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί αυτό το πλαίσιο. Εμείς μπορούμε να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο οποιαδήποτε χώρα θα ευεργετηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει και το θέμα ε, πληροφοριών για τους επιβάτες, το PNR, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να το συζητούμε με τους Αυστραλούς, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, έτσι ώστε η κίνηση προς τα έξω να είναι πιο ασφαλής, αλλά μας ενδιαφέρει και η εσωτερική ασφάλεια, δηλαδή στην ουσία θα είναι ασφαλέστερο να ταξιδεύει κανείς προς τις ΗΠΑ παρά από το Παρίσι στο Βερολίνο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση. Το σύστημα Eurodac θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο όλο σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα. Ως προς τα μέτρα κατά πολέμησης διαφθοράς, το ερώτημα Μακοβέη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Ουγγαρία ε, πέρασε ένας νόμος, εγκρίθηκε ένας νόμος που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας και θα θέλαμε να ε, λάβουμε υπόψη και την συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής των, ε, των υπεύθυνων για την πάταξη της τρομοκρατίας και τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λάβουν και να προωθήσουν. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Βλέπετε ότι ο Υπουργό για την κοινωνική ένταξη και ιδιαίτερα το θέμα της ένδειξης Ρωμά μας περιμένει με την ομάδα του εκεί και γι' αυτό τώρα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους βουλευτές που συνεργαστήκαν για να τελειώσουμε έγκαιρα και τέλος από κοινού να κάνουμε μια δήλωση κατά ε, καταδίκασε σε των ε, ε, φόνων και δολοφονιών που έγιναν χθε στη Μόσχα με 35 θύματα και πολλούς τραυματίες πρέπει από κοινού να δράσουμε κατά των τρομοκρατών και να προστατεύουμε τα θύματα τους. Τέλος θα θέλω να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Πιντέρ για την παρουσίασή του. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Θέλουμε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να ολοκληρώσουμε και να πραγματοποιήσουμε όλου του όρου που αναφέρθηκαν. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Dear colleagues, if you please be seated. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. We should kick off and get started because we got this. Λοιπόν, Πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολύ βαβαρημένο πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε την τιμή και ευχαρίστη να καλωσορίσουμε τον Υπουργό κοινωνική ένταξη τη Ουγγρική Προεδρία, που θέλει να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρία όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ένταξης και ειδικότερη ένταξη των Ρωμά. Ο κ. Ζολτάν Μπάλοκ, υφυπουργός για θέματα κοινωνικής ένταξης στην Ουγγαρία, είναι εδώ και θα έλεγα να προχωρήσουμε όπως κάναμε και προηγουμένως με τον πρώτα ένα γύρο ερωτήσεων για τους συντονιστές, το πολύ δύο λεπτά. Πρώτος γύρος αντιδράσεων του Υπουργού και κατόπιν ανοιχτό γύρο συζήτηση για να τελειώσουμε σε μια ώρα, μια ώρα και ένα τέταρτο το πολύ. Γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα για να ολοκληρώσουμε τα θέματα της μέσης διάταξης. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, είσαστε καλόδεκτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σήμερα συζητούμε μια προτεραιότητα έναν ε, τομέα για τον οποίο δεν είχαμε ιδιαίτερη εξωτερική πίεση για να τον θέσουμε ως ε, σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη της Προεδρίας της Ουγγαρίας. Το θέσαμε όμως ως προτεραιότητα εμείς με δική μας πρωτοβουλία. Ο λόγος ήταν ότι για πολλές δεκαετίες οι εμπειρογνώμονες προσπάθησε να καταλάβουν ή να λύσουν το πρόβλημα των Ρωμά στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ όμως η Ευρώπη δεν έχει δώσει την δέουσα προσοχή και σημασία στο θέμα αυτό, στην πολιτική της ατζέντα. Στους έξι μήνες λοιπόν της Προεδρίας μας θα θέλαμε να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Ο δικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια στρατηγική πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της ένταξης των Ρωμά. Και θα θέλαμε κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει και το δικό του εθνικό, τη δική του εθνική της στρατηγική ή τουλάχιστον να την προετοιμάσει για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο που εκπροσωπώ εγώ είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και εγώ είμαι υπεύθυνο για την κοινωνική ένταξη. Συζητούμε λοιπόν την ε, πλατφόρμα αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και της ένταξης ε, των Ρωμά, ε, της σχετικής στρατηγικής σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Οι περισσότεροι από εσά, οι αρκετοί από εσά είσαστε εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό και έχετε ενεργά αναφερθεί στο θέμα αυτό εδώ και καιρό. Πρέπει να ξέρετε ότι όντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν νέες ε, δηλώσεις ή να πει κάποιος κάτι καινούριο για το ζήτημα αυτό. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα έτσι ώστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Η δική μας εμπειρία στην Ουγγαρία δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνένεση, να υπάρξει μια θετική προσέγγιση, τουλάχιστον από την πλειοψηφία. η οποία συνήθως είναι ιδιαίτερως αρνητική για το θέμα των Ρωμά. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Βεβαίως πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα αυτό με σαφή, και με ξεκάθαρο τρόπο, έτσι ώστε να καταδείξουμε ότι αυτό το θέμα μας αφορά όλους και θα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με αυτό. Αυτό είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Μια άλλη πτυχή είναι το πώς αυτή η μειονότητα πώς ζει και πώς μπορεί να ενταχθεί και να βοηθήσει και η ίδια ενεργά στην επίλυση του προβλήματός της. Βεβαίω, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη λύση ως προς αυτό. Μπορεί να υπάρξει βεβαίως κάποια πρόοδο, αλλά δεν υπάρχει κάποια καθοριστική ε, λύση η οποία μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί και μάλλον θα ήταν και πολύ ε, φιλόδοξο να περιμένουμε ότι μέσα στο εξάμεινό μας θα υπάρξει λύση του προβλήματος αυτού. Οι κοινότητε των Ρωμά θα πρέπει να ε, μπλακούν, θα πρέπει να συμμετάσχουν, να δώσουν και οι ίδιες τη δική τους άποψη για τη στρατηγική που εκπονούμε, γιατί τους αφορά. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε ώστε να αναλάβουν και οι ίδιοι δράση είναι ανενεργοί, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ανεργία ή την έλλειψη προσόντων και δεξιοτήτων, αλλά δεν έχουν και την ε, ευκαιρία, αλλά ίσως και τη θέληση και οι ίδιοι να κάνουν κάτι. Αυτό λοιπόν εμείς θα θέλαμε να το ε, αντιμετωπίσουμε, θα θέλαμε να τους έχουμε ως ενεργούς συμμετέχοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. από την αρχή ήμασταν της ε, άποψης ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον της Ευρώπης, το θέμα των ε, Ρωμά. Μιλούμε για πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Βέβαια υπάρχουν ε, πάντα διαφορετικές απόψεις στο πώς είναι τελικά η Ρώμα, αλλά αν θεωρήσουμε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι 10 εκατομμύρια, είναι και άνεργοι και ε, αδύνατο να ενταχθούν στο ε, εργατικό δυναμικό. Υπάρχει τεράστια φτώχεια, υπάρχει μεγάλος κοινωνικός αποκλεισμός και αυτό βεβαίως είναι τυπικό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αν λοιπόν εμείς μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα είναι και ανθρωπιστική πράξη. Αλλά θα ικανοποιήσει και τα οικονομικά μας συμφέροντα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αλλά και οι κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει, ε, έχουν λάβει πολλές πρωτοβουλίες και έχουν δαπανίσει αρκετά χρήματα στα προγράμματα ένταξης των Ρωμά. Αλλά η κατάσταση των ίδιων των Ρωμά δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, μάλιστα έχει επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά τις συνθήκες ε, εργασίας και το επίπεδο διαβίωσής τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε και να το πούμε ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβεβαιώσει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές, η οικονομική και κοινωνική πληροφόρηση είναι και ενημέρωση είναι σημαντική για τα κρατημέλη. Είναι, για τα είναι θέμα σημαντικό και τα θεσμικά όργανα επίσης εδώ πρέπει να παίξουν τον ρόλο που του αναλογεί. Πολλέ έρευνες έχουν δείξει ότι η ένταξη των Ρωμά δεν είναι απλώς μια ανθρωπιστική πράξη αλλά και οικονομική πράξη γιατί ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, ε, τη βιωσιμότητα των ε, ε, συστημάτων κοινωνική πρόνοια. Οπότε η ένταξη των Ρωμά είναι πραγματικά υψίστη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημοσιευθεί μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εάν ο βαθμός απασχολησιμότητας των Ρωμά έφτανε το περιφερειακό, τον περιφερειακό μεσόωρο, τότε το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 46%. Αυτό είναι τεράστιο νούμερο και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και από κοινωνικής αλλά και από α, οικονομικής πλευράς. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε το θέμα της εκπαίδευσης, της στέγασης, της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης, της υγείας. Πρέπει όλους αυτούς τους τομείς να τους δούμε με έναν συνολικό και συνεκτικό τρόπο. Πρέπει να τους δούμε παράλληλα η ε, Ουγγρική Προεδρία ελπίζει να υπάρξει κάποια πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ένταξη των Ρωμά. Βεβαίω πρέπει να γνωρίζετε ε, αυτά τα γεγονότα, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία ήδη, αλλά ε, εγώ είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος που η τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, από την Ουγγαρία ξεκίνησαν μια τέτοια πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι τον Φλεβάρι του 2011 θα μπορέσει να εγκριθεί η σχετική έκθεση που προέκυψε. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει και την Κομισιόν αλλά και το Συμβούλιο στην δουλειά που έχουν να κάνουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 6 Απριλίου του 2011 θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα των κρατών μελών, το στρατηγικό πλαίσιο για την ένταξη των ρωμάς, το πρώτο σχέδιο βέβαια, και θα εγκριθεί ε, από το Συμβούλιο επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας. Στο τέλος της ε, Προεδρίας μας θα θέλαμε να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει το σχέδιο αυτό και βεβαίως ε, θα παρακολουθούμε και εμείς στενά τις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ. Υπάρχει μια ομάδα κρούσης, μια task force, η οποία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη πέρσι και ασχολήθηκε με ένα ε, ε, ερωτηματολόγιο μέχρι το Δεκέμβρη, το οποίο ερωτηματολόγιο απεστάλλει στα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα είναι το καθήλυν αρμόδιο ε, συμβούλιο για τις συζητήσεις περί των συμπερασμάτων. Βεβαίως θα συμπεριληφθούν και οι απόψεις άλλων συμβουλίων, όπως ας πούμε το Συμβούλιο ε, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και νεολαία, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επίσης θα συζητήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία ελπίζουμε μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να μπορούν να εγκριθούν. Θα θέλαμε λοιπόν να, μέχρι τότε να μπορεί να γίνει αυτό, να μπορούν να εγκριθούν τα συμπεράσματα. Οι βασικές πτυχές των συμπερασμάτων του Συμβουλίου θα είναι οι εξή θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, καταγράψουμε δεσμεύσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι τομείς παρέμβασης με συγκεκριμένους δείκτες και ποσοτικούς στόχους. Πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένους στόχους αλλά όχι αποκλειστικού. Όταν λοιπόν καθορίσουμε μια ομάδα στόχων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα ε, εδαφικά και εδαφικές πτυχές αλλά και κοινωνικές. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση την, ε, ε, του μέλους του, του Ευρωβουλευτού Γιαρούκο για το συγκεκριμένο αυτό ε, θέμα όπου, θα, όπου προτείνει να δημιουργηθεί ένας χάρτης που θα περιλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες περιοχές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις κυβερνήσεις στην εκπόνηση των δικών τους σχεδίων ελέγχου και καταγραφής αλλά και εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνδέσουμε το θέμα της ένταξης των Ρωμά με τις υπόλοιπες πολιτικές έτσι ώστε όταν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία να είναι σαφώς συνδεδεμένη η στρατηγική για τους Ρωμά με την στρατηγική για το 2020. ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένε δεσμεύσει λοιπόν για την, ε, για την ε, πολιτική για του Ρώμα ω τμήμα τη στρατηγική για το 2020. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένου δείκτες καθώ επίση και ποσοτικούς στόχου στα εθνικά τους προγράμματα έτσι ώστε να προωθήσουν την, ε, την απασχόληση και να μειώσουν την, τον αποκλεισμό που υφίστανται οι Ρωμά. Για να είμαστε λοιπόν επιτυχή σε αυτό μας το εγχείρημα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, και τα έγγραφα τα οποία ορίζουν αυτές τις δράσεις και, και να μπορέσουμε να, τα, να συντονιστούμε με, και, με, και σε διεθνές και σε ε, τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το εργαλείο, το μέσο για να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές, τους ε, ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς πόρους. Θα θέλαμε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το γεωργικής ανάπτυξης και ανάπτυξη υπαίθρου. Ε, θέλουμε λοιπόν να συντονιστούν όλα αυτά τα ταμεία έτσι ώστε να υπάρξουν συνέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε βιώσιμη πολυετή, βιώσιμα πολυετή και μακροπρόθεσμα προγράμματα. Όσοι λοιπόν ε, εργάζονται επί τόπου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως δημιουργείται έτσι ένας κάποιος πανικός για το τι γίνεται όταν πάβουν να υπάρχουν κονδύλια. Γι' αυτό ε, προτείνουμε αυτό τον, αυτό τον κατάλογο δικτών ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, παρακολούθηση. Πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, αυξημένη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την πρόσβαση στα κονδύλια και σε σχέση με το πώς προωθούνται οι διάφοροι διαγωνισμοί για την προσφορά βοήθεια σε, τέτοιους, σε τέτοιες μειονεκτούσες ε, κοινωνικές ομάδες. Ε, βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις για το θέμα αυτό ευχαρίστω να σας απαντήσω αλλά συνοπτικά μπορώ να πω ότι αυτά τα τρία ζητήματα η ε, παιδική ε, φτώχεια, η φτώχεια αλλά και η, συμπερίληψη των, ε, η ένταξη των Ρωμά είναι θέματα τα οποία θα δείξουν κατά πόσο είμαστε αξιόπιστοι. Πριν από 20 χρόνια, όταν σταμάτησε η δικτατορία στην Ουγγαρία, εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό κράτος και ένα κράτος ασφαλές, αλλά τώρα κάποιοι λένε ότι καλύτερα ήταν όταν είχαμε δικτατορία παρά τώρα που έχουμε δημοκρατία σε ό,τι αφορά την, ε, τα κοινωνικά θέματα. Οπότε για μας είναι σημαντικό να επιτύχουμε έτσι ώστε να δείξουμε ότι η δημοκρατία έχει ισχύ και να δείξουμε ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε για αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που δεν είναι σε θέση να υποφεληθούν ε, της δημοκρατίας και της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως μπορούμε εμείς. Αυτή είναι λοιπόν η ε, η ψυχολογική διάσταση, αν θέλετε, τη ένταξη των ε, Ρώμα και τη αντιμετώπισης της φτώχειας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ε, συντονιστές εκ των προτέρων, διότι θα αρκεστούν στα δύο λεπτά. Ο κύριος Σόγκορ έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Ουγγρική Προεδρία διότι αναλαμβάνει αυτό το θέμα και του προσδίδει τη σωστή του σημασία. Γνωρίζουμε ότι στην Ουγγαρία υπάρχει ένα Υπουργείο που ασχολείται ειδικά με αυτά τα 10-12 εκατομμύρια Ρωμά που ζουν κάτω από ε, πολύ και κακές συνθήκες, συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Υπάρχουν πολλοί ε, Ρωμά που ντρέπονται να, αναφέρουν, να αναφέρθουν στην εθνότητά τους. Και οι πόροι είναι ανεπαρκείς έτσι κι αλλιώς για να τους καλύψουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επινοηθούν διαφορετικά τα προγράμματα ε, έτσι ώστε οι Ρωμά να μην ε, έχουν αυτό το αίσθημα ντροπή. Θα ήθελα να πω το εξής ως προς την εφαρμογή του νόμου. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι γνωστό το θέμα του ολοκαυτώματος των Ρωμά. Στην χώρα μου, στη Ρουμανία, υπήρξαν, έγιναν πόγκρομ και κατά τη δεκαετία το Μάρτιο του 1990 όπου έγιναν πολλές συγκρούσεις και δυστυχώς συνελήφθηκαν μόνο ακτιβιστές Ρωμά. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά είδη ολοκαυτώματος. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, πρωτοβουλία και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Η κυρία Μπόσκουρτ από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτή την παρουσίαση. Είσαστε πολύ φιλόδοξος και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Θέλετε να φτάσετε σε έμπρακτες λύσεις κατά την Προεδρία σας Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να εκπονήσετε μία στρατηγική η οποία να μην προβαίνει μόνο σε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Πώς θέλετε να προωθήσετε περαιτέρω το όλο ζήτημα και έμπρακτα ποια μέτρα θα λάβετε μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Είπατε ότι έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα αλλά Μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί στην Ουγγαρία, πώς αντιμετωπίζει η ίδια η Ουγγαρία αυτό το θέμα μέχρι τώρα. Πώς ε, αντιμετωπίζετε μια συνολική σφαιρική στρατηγική. Νομίζω ότι μιλήσατε για ένα ειδικό ε, project. Τι πιστεύετε ως προς την ύπαρξη ενός ενιαίου κέντρου αποτίμησης. Θα πρέπει να έχουμε μία οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα στην Ευρώπη και τι, θα, τι προτίθεστε να κάνετε κατά την Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ από τους Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Από το Κοινοβούλιο έχουμε αποστείλει διάφορα μηνύματα. Θα θέλαμε δηλαδή να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια ε, προσέγγιση πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια θα ήταν η νομική βάση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να δεσμεύονται να εγκρίνουν τέτοιες εθνικές στρατηγικές. Γιατί αν δεν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο, πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κρίσης. Τι θα γίνει αν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, ποια θα ήταν η νομική βάση έτσι ώστε να υπάρχει υποχρεωτικό συντονισμός των ε, χρημάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μιλήσατε για το 2020. Από τη δική σας πείρα στην Ουγγαρία, τα τελευταία 20 χρόνια. Πιστεύετε ότι 8 με 9 χρόνια αρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επίσης, επειδή ασχολείστε με θέματα κοινωνικής ε, ένταξης, αυτό είναι ένα άλλο από τα χαρτοφυλάκια σας, μιλήσατε για την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψη της Ουγγρικής ε, Προεδρίας για την ε, καταπολέμηση της διάκρισης με βάση το φύλλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ευχαριστώ από ε, Γκουέ, κυρία Έμστεν. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την κατάσταση των ΛΟΜΑ στην Ευρώπη, ξέρουμε πολλά νομίζω τώρα πια. Δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε όλα και τα εμβαθύνουμε. Θα πρέπει να καταλήξουμε επιτέλους σε συμπεράσματα. Οι ερωτήσεις που είναι εξή. Πρώτον, δεν νομίζω θα ωφελήσει αν εκ μιας αρχής ε, συμμεληφθούν οι Ρώμα στις αποφάσεις που θα λεφθούν για αυτούς. Πώς θα το πραγματοποιήσετε αυτό στα συμπεράσματα που θα προετοιμαστούν και θα αποδηγήσουν στην απόφαση του Συμβουλίου. Δηλαδή, δεσμευτική συμμετοχή των Ρωμά. Ποιε είναι οι δομέ που θα δημιουργηθούν για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, αναφερθήκαν οι κοινοτικοί πόροι. Υπήρξαν επαρκεί πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα τελευταία χρόνια και δεν το ε, χρησιμοποίησαν τα κράτα-μέλη Πώς θα φροντίσετε αυτοί οι πόροι πραγματικά να απορροφηθούν. Πώς θα φροντίσετε να διευκολύνετε την ε, πρόσβαση οργανώσεων των Ρωμά στα κράτη-μέλη ή να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, αυτά τα, ε, αυτά τα χρήματα. πιο είναι ο του, κοινωνικού ταμείου, του κοινωνικού κοινοτικού ταμείου. Συγγνώμη. Τρίτον, τα μέτρα που θα ληφθούν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του αντιτσιγκανισμού ποια θα είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω γιατί αν δεν υπάρχει πραγματική παρέμβαση και κρατική εδώ όλες οι προσπάθειές μας δεν θα καρποφορήσουν Τέλος, αναφερθήκατε στην ένδια παιδιών σε σχέση με τη στρατηγική για τους Ρωμά. Ποιος είναι ο ρόλος που θα δώσετε εδώ στην παιδεία. Όσον αφορά δηλαδή την παιδεία, τι θα συμπεριλάβετε από το τομέα αυτό στη στρατηγική για τους Ρωμά. Μου φαίνεται πάρα πολύ κεντρικό το σημείο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ΣΥΑΡ, όχι, μην είναι γεγραμμένη. Η κυρία Μόρμπα, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα τη δική μου εμπειρία, η Ρωμά και οι πιο ευάλωτοι, τα παιδιά δηλαδή και οι γυναίκες, υποφέρουν από βία μέσα στις δικές τους κοινωνίες. το κράτος εκάστοτε δεν τους υποστηρίζει λόγω κάποιος κακά εννοούμενης ε, πολιτικής ορθότητας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εθελοτυφλούμε παραδείγματος χάρη σχετικά με την πορνεία που αφορά νέες κοπέλες Ρωμά που δεν τους επιτρέπεται καν να πάνε στο σχολείο. Γιατί λέγεται ότι τα κορίτσια των Ρωμά πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στο σχολείο, να ασχολούνται με τα μικρά τους αδέλφια κλπ. Πρόκειται να κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη μορφή της ε, καταπίεσης και της διάκρισης εις βάρος ενός ε, φίλου. Κάτι άλλο που είναι ένα πρόβλημα για την ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία ε, το πρόβλημα είναι οι ψηλά επιτόκια που επιβάλλουν διάφοροι τοκογλήφοι στους Ρωμά. Αυτό δεν επιτρέπεται και εμένα μου έρχονται στα χέρια μου πολλές εκατοντάδες επιστολών από ουγγρικές ε, ε, οικογένειες Ρωμά που λένε ότι οι όροι τους οποίους είναι αναγκασμένοι να ζουν είναι παρόμοιοι με εκείνους στον τρίτο κόσμο γιατί τους επιβάλλονται αυτά που δηλαδή βρωμιά, έλλειψη υγιεινής, πράγμα που δεν θέλουν να δεχθούν. Και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολλές νομότυπες οικογένειες Ρωμά που ενοχλούνται από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν. Τρίτος κόσμος. Το κράτος δεν δρά. Και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση μέσα στα πηγές της κοινοτικής στρατηγικής Ρωμά θα πρέπει να ανυποθετηθούν αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να αντιδράσετε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας και για να απαντήσω προς τον κύριο Σόγκορ. Θα ήθελα να πω ότι τα σχόλιά του ήταν ιδιαίτερα σημαντικά Υπάρχει λόγος ε, που ονομάσαμε το Υπουργείο θέμα ε, ένταξης, κοινωνικής ένταξης και δεν μιλήσαμε για ένταξη των Ρωμά αποκλειστικά. Μπορώ να σας δώσω πολλά ε, παραδείγματα από την Ουγγαρία. Θα μπορούσα να σας δώσω και αριθμητικά στοιχεία για ολόκληρη την Ευρώπη. Το 80% ε, των Ρωμά ζουν από, κάτω από συνθήκες απόλυτης φτώχειας και το 20% βρίσκεται στην Ουγγαρία. Η φτώχεια δεν είναι προνόμιο των Ρωμά, αλλά προνόμιο και δυστυχώς και άλλων εθνοτήτων. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία κοινωνική προσέγγιση και όχι εθνοτική. Όποιος είναι κάτω από το κατόφλι της φτώχειας θα πρέπει να έχει κάποιας μορφής αρρωγή. Και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τους ε, Ρωμά. Ε, τέθηκε θέμα καταπολέμησης των διακρίσεων. Νομίζω ότι πολλές φορές οι διακρίσεις βασίζονται στην εθνότητα. Θα πρέπει όμως να έχουμε μία συνολική στρατηγική που να βασίζεται σε μια κοινωνικού χαρακτήρα προσέγγιση. Θα πρέπει να δώσουμε τέλος στην φτώχεια. Επίσης, ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε είναι η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα ήθελα να πω ότι στην Ουγγαρία, 400 χρόνια πριν, η, διορίστηκε πρώτη κυβέρνηση αντιμετώπιση του θέματος τον Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μία μακραίωνη παράδοση. Αλλά αν υποβάλουμε το ερώτημα πώς ορίζεται ένας Ρωμά σήμερα, δεν είναι εύκολο να δώσουμε ε, μία απάντηση. Βεβαίως έχει σημασία να δηλώνονται όλοι οι Ρωμά, δεν το κάνουν πάντα. Κατά την τελευταία απογραφή το 190.000 δηλώθηκαν ως Ρωμά. Αν δείτε όμως τα ε, στοιχεία που μας έδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, μιλούν για 780.000 Ρωμά. Και υπάρχει ένα αίσθημα κατά των Ρωμά. Εκεί γίνεται λόγος για 1,5 με 2 εκατομμύρια Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε αυτές τις ομάδες, ποιες είναι οι ομάδες ε, στόχοι. Επίσης ε, μας ε, απασχόλησε αυτό το θέμα, δηλαδή κατά πόσο θα πρέπει να βασιστούμε στην εθνότητα καθαρά. Αυτό που έχει σημασία είναι η χρήση των πόρων. Χρειάζεται να κάνουμε ένα πολύ σωστό βήμα προς το εμπρός και θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ένας κοινοτικός οργανισμός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα, δηλαδή να προβάλλουμε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με μία εθνοτική καθαρά ομάδα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ευεργετούνται αυτές οι ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχονται αυτά τα στοιχεία με μία ανώνυμη βάση δεδομένων. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να μετρήσει τα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά τα προγράμματα φτάσαν στους Ρωμά ή όχι. Γιατί πολλοί λένε ότι αν ε, τα χρήματα πάνε στους Ρωμά, τότε όλοι δηλώνονται ως Ρωμά, ενώ αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο δεν έχει λόγο να το δηλώσει κανείς. Αυτό είναι κάτι το αυταπόδεικτο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ελέγχουμε τη, τους όρους ε, υποβολής αλλά και την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων, εάν είναι αποδοτικά ή όχι. Εάν λοιπόν κάποιος έχει πληγή, ε, πληγεί, το Τέργου αναφέρθηκε για τη δεκαετία του 90, αλλά έγιναν και άλλα πογκρόμ ανά τους αιώνες. Γι' αυτό θα πρέπει για ιστορικούς λόγους η δικαιοσύνη να αναλάβει αυτό το έργο. Η κυρία Μπόσκουρτ μου μίλησε για την ε, πραγματιστική μας προσέγγιση, για την έμπρακτη προσέγγιση. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές, αλλά Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από συστάσεις και υποδείξεις αυτή τη στιγμή. Πιστεύω όμως ότι τη στιγμή που το Συμβούλιο θα έχει ε, εγκρίνει αυτά τα συμπεράσματα και όταν έχουμε πληροφορίες πιστεύω ότι θα δούμε γιατί τα προγράμματα κατά των διακρίσεων δεν ήταν τόσο αποδοτικά. Ελπίζω όλα αυτά να έχουν επίπτωση στα κράτη-μέλη, να απασχοληθούν και τα κράτη-μέλη και να δουν γιατί δεν φτάσαμε στην επίτευξη των στόχων μέχρι τούδε. Δεν ξέρω κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό θα επιτύχει. Μιλάμε για βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει όμως να μιλάμε για κακές ή χειρότερες πρακτικές θα πρέπει να καταρτήσουμε και τέτοιους αρνητικούς καταλόγους, διότι πολλές φορές μαθαίνουμε πολύ περισσότερα από τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να έχουμε και αρνητικούς καταλόγους, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα που δεν ήταν αποδοτικά, ιδιαίτερα όταν τα κονδύλια δεν πάνε στους σωστούς ανθρώπους. Κυρία Βέμπερ, ρωτήσατε γιατί δεν είναι ευρωπαϊκή αυτή η στρατηγική γιατί δεν μιλάμε για ένα πλαίσιο εθνικών ε, στρατηγικών. Πρόκειται για έναν επιμερισμό εργασίας. Τα κράτη-μέλη φέρουν τη δική τους ευθύνη, την εθνική ευθύνη και υπάρχει και η ευρωπαϊκή παράλληλα. Και εδώ εντάσσεται και η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτά τα 8, 9, 10 χρόνια που έχουμε μέχρι το 2020 δεν θα αρκέσουν για να βρούμε μια λύση, αλλά τουλάχιστον να αναχαιτήσουμε την επιδίνωση. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι μια επονίδιστη κατάσταση εδώ και 20 χρόνια η κατάσταση των Ρωμά επιδεινώθηκε, δεν βελτιώθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια αρνητική τάση που διαγράφεται, δηλαδή αυτοί που ζουν κάτω από κατάσταση απόλυτης φτώχειας δεν είδανε καμία βελτίωση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε επίσης και τις διακρίσεις. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο όταν ε, έρχονται, φτάνουν οι αστυνομικέ δυνάμεις, τότε κανένας δεν εμφανίζεται ως Ρωμά. Και αυτό φαίνεται από την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το αρνητικό συνέστημα και οι άνθρωποι θεωρούν ότι όταν προσέρχεται η αστυνομία καλύτερα να μην δηλωθώ ως Ρωμά διότι τότε θα έχω ε, διπλό πρόστιμο ή θα είμαι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Ο κύριος Πίντερ μίλησε για ένα διτό ε, πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την αστυνομία, έτσι ώστε οι αστυνομικές ε, δυνάμεις να μάθουν να δρουν σωστά, να μεταχειρίζονται δίκαια, να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση των ε, Ρωμά και να αντιμετωπίζουν σωστά και το έγκλημα, την αντιμετώπιση του εγκλήματος ως προς την εθνοτική προσέγγιση. Υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο θα σταθούμε ιδιαίτερα επιτυχής. Δηλαδή, έχει σημασία να αυξηθούν και οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά θα πρέπει οι Ρωμά να ενταχθούν και στο σχολείο, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να εκπαιδευτούν ως αστυνομικοί. Ίσως και αυτό θα βοηθούσε στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Δηλαδή αν έχουμε μία μέση τάξη Ρωμά σε ένα κράτος μέλος αυτό θα ήταν ιδιαίτερα θετικό. Και ήδη έχει επιτελεστεί κάποια πρόοδος. Υπάρχει και ένα λόμπι Ρωμά Άρα υπάρχει εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει σημασία όμως η κατάρτισή τους έτσι ώστε να γίνουν μηχανικοί, γιατροί και ούτω καθεξής. Θα βοηθούσε το εθνοτικό ζήτημα. Ως προς το ε, ερώτημα της κυρίας Έρνστ, είπα ότι πράγματι αυτό θα είναι ένα βήμα αποφασιστικής σημασίας. Όταν κάποιος είναι υποκείμενο και όχι αντικείμενο ενός μέτρου και όταν κάποιος αναλαμβάνει δράση, είναι δηλαδή ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας, έχει μία διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Εμείς προσδίδουμε μεγάλο, ε, μεγάλη σημασία στην πολιτισμική ταυτότητα των Ρωμά. Χωρίς πολιτισμική ταυτότητα δεν μπορεί κανείς να ανέλθει το, τα κοινωνικά κλιμάκια αν δεν εντάσσεται σε μια κοινότητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία για τους Ρωμά. Άρα δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα, πρέπει να μάθουμε την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους καλύτερα. Στην ε, Ουγγαρία υπάρχουν ε, και βιβλία ρωμαλογίας. Μιλάμε για, ασχολούμαστε με την παράδοσή τους, υπάρχει ένα ειδικό μάθημα στα σχολεία και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο δράσης όπου οι Ρωμάνα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα στην Ουγγαρία, αλλά δεν είναι πάντα ε, επαρκώς λειτουργικό. Υπάρχουν πολλά, αρκετά συμβούλια των Ρωμά και υπάρχουν πέντε πολιτικοί που εκπροσωπούν την κοινότητα αυτή από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη. Ε, εκλέγονται άμεσα οι εκπρόσωποι αυτοί και υπάρχει και μία εθνική, ένα Συμβούλιο Εθνικής μειονότητας με 53 μέλη εξέλιξαν τον πρόεδρό τους την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα αυτό το σύστημα φτάνει και στο μικρότερο χωριό όπου διαβιούν Ρωμά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, Ρωμά έτσι ώστε να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τα πραγματικά τους συμφέροντα Πήγα και στη Ρουμανία την προηγούμενη εβδομάδα, είδα πώς εκπροσωπούνται οι Ρωμά σε πολιτικά φόρα και άλλα φόρα και είναι δύσκολο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. αν δεν λάβουμε υπόψη και την περιφερειακή εκπροσώπηση. Πολλές φορές δεν χρησιμοποιήθηκαν και τα κοινοτικά κονδύλια επαρκώς. Θα ήθελα αυτό να ενταχθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Άρα όταν προκυρήσετε ένας ε, διαγωνισμός θα πρέπει να γίνεται κατανοητός από όλους, διότι υπάρχουν 770 ε, υποδιαιρέσεις και μάλλον ε, διαχωρισμένες περιφέρειες όπου διαβιούν Ρωμά. Και η προηγούμενη Ουγγρική κυβέρνηση προκήρυξε διαγωνισμούς όπου μία μόνο κοινότητα υπέβαλε αίτηση και μετά απέσυραν την αίτησή τους. Άρα ποιος φταίει, φταίει η κυβέρνηση και ίσως η διατύπωση είναι προβληματική και ίσως ε, ιδιαίτερα δυσνόητη. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το σύστημα. Μιλήσατε και για την καταπολέμηση αυτού του αισθήματο κατά τον ε, Ρωμά. Αυτό το είπα όταν μίλησα και για την αστυνομία και την αντιμετώπιση της αστυνομίας θα πρέπει να είμαστε να συζητάμε τα θέματα των ε, Ρωμά και τα σχετικά προβλήματα. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε τα αρνητικά αισθήματα έναντι των Ρωμά. Μίλησα για το μάθημα της ρωμαλογίας και είπα ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτήν την κοινότητα καλύτερα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το μάθημα στο σχολείο. Θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Έγινε λόγος και για την, φτώχεια, την παιδική φτώχεια. Υπάρχει μία ευρωπαϊκή στρατηγική επί του θέματος και για την Βελγική Προεδρία φτάσαμε σε πολύ καλά συμπεράσματα. Μιλήσαμε για το ότι θα πρέπει τα παιδιά να τα δεχόμαστε σε βρεφονιπιακούς σταθμούς από πολύ μικρή ηλικία, στα νηπιαγωγεία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και έτσι μόνο θα μπορέσουν να ενταχθούν και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να πω στην κυρία Μορβάη ότι αν δεν είχατε μία εθνοτική προσέγγιση θα συμφωνούσα μαζί σας. Εάν δείτε ποιοι ζουν κάτω από ε, μία κατάσταση απόλυτης φτώχειας, πρόκειται για ένα τραγικό φαινόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για την ε, καλύτερη για την βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, δηλαδή πουλούν τα παιδιά τους ή τα εκδίδουν. Γνωρίζετε ότι αυτό το φαινόμενο δεν σχετίζεται μόνο με τους Ρωμά. Αν ε, βρεθείτε στο Άμστερνταμ σε ορισμένους δρόμους, βλέπετε ότι υπάρχουν και νέες γυναίκες από την Ουγγρα... Ουγγαρία που εργάζονται, που εκδίδονται. Μερικές δεν ε, είναι Ρωμά. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι εγκλήματος που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους και χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένη δράση. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά εθνοτικό λοιπόν το ζήτημα. Είναι κάτι που σχετίζεται με την φτώχεια. Αυτά είχα να πω εν ολίγης. Thank you. Thank you for the Ευχαριστώ πολύ για τις ενδράσεις σας και τις πολύ προσεκτικές απαντήσεις που δέχεται σε κάθε σημείο. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε ένα νέο γύρο ερωτήσεων. Έχω ένα μακρύ κατάλογο. Οκτώ. Οκτώ. Μελή. Θα σας διαβάσω και θα κλείσει μετά ο κατάλογος. Mrs. Guillaume, Mr. Ensue, Mr. Brons, Mrs. Infeld, Mr. Marinescu, and Mr. or Mrs. Mrs. Yotova. Yotova. Αλλά βλέπω ότι η κυρία Μπότσκουρτ θέλει να κάνει μια παρατήρηση διαδικαστική ίσως. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση για την οριζόντια οδηγία. Η συνάδελφος Βέμπερ υπέβαλε την ίδια ερώτηση και δεν πήραμε απάντηση. Είμαι σίγουρο ότι παραβλέφθηκε, αλλά θα ήταν καλό να ακούσουμε κάτι σχετικό. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε, να είστε πιο συγκεκριμένος για την οριζόντια οδηγία. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Αυτό δεν είναι απαραίτητο τμήμα του προγράμματος Προεδρίας. Δεν έχω νέες πληροφορίες για το θέμα. Δεν το ξέχασα ότι υποβάλλει την ερώτηση, αλλά δεν είχα τίποτα στην πραγματικό να σας πω. Ωραία, περάσαμε στο δεύτερο γύρο τώρα. Τέλει και άλλο σχόλιο. Ναι, υπήρχε ίσως μια ε, παρεξήγηση. Α, εσείς αναφερθήκατε οριζόντια οδηγία, οδη, αναφερόσαστε στην οδηγία κατά των διακρίσεων. Α, στην προκειμένη περίπτωση έχω να σας απαντήσω διαφορετικά. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας να την μεταφέρουν στον εθνικό δίκαιο και να την εφαρμόσουν. Δεν είναι θέμα της ε, Προεδρίας. Ε, Πρόεδρος, μα υπάρχει μια νέα οδηγία που ακόμα δεν έχει εγκριθεί Akkor a harmadik kísérlet, Κοίταξτε, μπορώ να αναβάλω την απάντηση απάντηση. Θα κάνω μια τρίτη προσπάθεια. Δεν είχα καταλάβει. Πραγματικά ήταν μια παρεξήγηση γιατί είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό. Ένα άλλο Υπουργείο είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα και η οδηγία αυτή έχει σαν στόχο τους αναπήρους και το θέμα του σεξουαλικού προανασταλισμού της διακρίσης βάση θρησκείας και από όσο ξέρω όσον αφορά τους αναπήρους και τα άτομα με ανάγκες θα υπάρχει κάποια πρόοδο στην ε, οδηγία αλλά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και γι' αυτό δίστασα να σας απαντήσω. Δεν ξέρω τώρα αν θα σας βοηθήσει η απάντηση που σας έδωσα. Πρόεδρος, καλά θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ο καθένας και να έχουμε μια τελική απάντηση από τον Υπουργό. Κυρία Κάντς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, εδώ θα πούμε ότι το θέμα της, ε, των διακρίσεων θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα εξαλειφθεί όχι μόνο στον τόπο εργασίας αλλά και σχετικά με τη θρησκεία, τον ε, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Ένα θέμα που αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει στο Συμβούλιο και γι' αυτό θέλαμε η Ουγγαρία προεδρεύουσα του Συμβουλίου να προωθήσει το θέμα. Θα είναι πολύ μεγάλη σημασία. Και για το δικό σας τον τομέα, δηλαδή για την ένταξη των Ρωμά. Γιατί πρόκειται για μια ε, η περίπτωση διακρίσεων και εδώ και γι' αυτό η έλλειψη των διακρίσεων δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στον χώρο εργασίας. Η δική μου ερώτηση αναφέρεται στην ε, φτώχεια των παιδιών και στην άνηση μεταχείριση πολύ κεντρικό το θέμα αυτό. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την ε, παιδεία ε, να διαχωρίζονται τα παιδιά κατά στο σχολείο ή όχι. Αυτό συζητιέται στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Επίσης το θέμα του συστήματος προσωπικού εισοδήματος ε, συζητιέται επίσης στην Ουγγαρία και ευνοεί αυτό τις πιο ε, πλούσιες οικογένειες. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Γκυλιόμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βέβαια το θέμα παρουσιάστηκε ευρέως ε, και στην αρχή αυτών που είπατε και που είναι σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις της ε, Προεδρίας για τους Ρωμά. Αναφερθήκατε στη τραγική πλαίσιο Είναι σαφές νομίζω ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ε, εφαρμόζεται στα ε, χώρα προέρευσης αλλά και στα χώρα, α, στις χώρες άφηξης. Το θέμα της ένταξης των δομά γενικά ετέθη ήδη και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο μπορείτε να ε, διευκρινίσετε κάποια θέμα όσον αφορά τις χώρες προέλευσης και τις χώρες ε, αποστολής αν θέλετε εξάρτησης των Ρώμα. Ποιοι είναι επίσης οι στόχοι της Ουγγρικής Προεδρίας ούτως ώστε η κοινωνία των πολιτών των Ρωμά να ενταχθεί στην ε, ε, ενέβρεση μιας λύσης για τις ομάδες αυτές, για τους Ρωμά δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σέλσιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία που συμπερέλαβε τα προβλήματα αυτά στις προτεραιότητες της. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά λίγο κάτι που ρώτησε και η συνάδελφος και κατόπιν όσον αφορά την μελλοντική στρατηγική πλαίσιο για τους Ρωμά, για την Ένωση Ρωμά θα είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική ή θα είναι μια συνάθρηση των επιμέρους κρατικών πολιτικών. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή και συνεπής πολιτική όσον αφορά τους Ρωμά και για το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη μέρη στα οποία θέλουν να εγκατασταθούν οι Ρωμά άσχετα από το που προέρχονται. Δεύτερον, θα ήσασταν υπέρ της εφαρμογής προγραμμάτων για τους Ρωμά μόνο μέσω των ε, τοπικών αρχών. Θέλετε δηλαδή μόνο οι τοπικές αρχές να είναι εκείνες που θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα μια που εκείνες ξέρουν τα επιτόπου προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Γκάλ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. ε, ικανοποίηση σα ήταν να ερχόσαστε εδώ και να μπορούμε να σα υποδεχθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί μέχρι στιγμή η σταδιοδρομία σα. πραγματικά ήταν σύμφωνη με τα προβλήματα που μας αναφέρετε εδώ μέσα στα πλαίσια της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρόσφατα συζητήσαμε πολλά οικονομικά θέματα και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας είναι επαρκείς για να επιτευχθούν οι στόχοι ή χρειάζονται συμπληρωματικοί πόροι για να μπορέσει η πολιτική αυτή να γίνει λειτουργική. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ. Η κυρία Εντφέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονό ότι η Ουγγρική Προεδρία έθεσε το θέμα αυτό ψηλά ε, στο πρόγραμμά της ε, και στις προτεραιότητες και βλέπω ότι δεν διστάστε να αναφέρετε διάφορες ε, διακριτικές μεταχειρήσεις και πρακτικές. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέμα βέβαια πολιτικής βούλησης και δεν ξέρω κατά πόσον όταν εφαρμόσουμε την πολιτική της ένταξης των Ρωμά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ορισμένες χώρες μέλη είναι κάπως θεσμοποιημένη αυτή η διάκριση και υπάρχουν και μαζικές διώξεις παρόλο που δεν το λέμε, δεν τις αποκαλούμε έτσι. Και υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσεις που δεν υποστηρίζουν τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε. Δεν κατάλαβα, το δικό σας Υπουργείο δεν είναι υπεύθυνο γενικά για τα μέτρα ε, υπέρ της καταπολέμησης των διακρίσεων γιατί πιστεύω ότι η νέα αυτή οδηγία που εκκρεμεί από το Συμβουλίο θα πρέπει να προωθηθεί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι όσον αφορά μία πάρα πολύ ε, αρνητική ρήτρα στο νέο σας νομοσχέδιο για, το, για τα ΜΜΕ αλλά ξέρω ότι κατάλαβα δεν είναι αρμόδιο το δικό σας υπουργείο γι' αυτό. Δεν ξέρω ότι η Προεδρία θα προωθέσει και το θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων κατά των ομοφιλοφίλων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ που μεταξύ των προτεραιοτήτων της Προεδρίας θα συμπεριλάβατε και το θέμα αυτό της στρατηγικής ε, υπέρ των Ρωμά. Ελπίζω να καταφέρετε να καταλήξετε σε μια ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μόνο μια εθνική. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και σχέδια που μπορούν να εφαρμόσουν στα κράτη-μέλη, ταυτόχρονα όμως με μια ευρωπαϊκή διάσταση. Και για να επανέλθω σε κάτι που είπατε, δηλαδή ελάχιστο αριθμό ε, θέσεων στα σχολεία ή και στις ε, αστυνομικές ακαδημίες για τους Ρωμά όλα αυτά μου φαίνεται ότι είναι σημαντικά υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα στη Ρουμανία και θα ήταν νομίζω καλό να το συμπεριλάβουμε γενικά στην ε, πολιτική υπέρ των Ρωμά η πλειοψηφία των Ρωμά είναι φτωχή και οπωσδήποτε αυτή η φτώχεια από ό,τι φαίνεται σχετίζεται με την ανεργία η ανεργία σχετίζεται με την έλλειψη ε, προσόντων και ικανοτήτων που θα βοηθούσαν στην εξέβριση της εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε κυρίως την παιδεία. Μόνο αυτή θα επιτρέψει να μπορέσει να υπάρχει μακροπρόθεσμα πρόοδος. Ελπίζω λοιπόν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιτρέψουν τα παιδιά Ρωμά να ενταχθούν στα σχολεία θα πρέπει να προωθηθούν θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίως για το Ρωμά που μετατίθεται από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτέ είναι μόνο προτάσει που θέλω να κάνω, όχι οριστήσει και ελπίζω να τι λάβετε υπόψη για τι επιδικίες σα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που συμμετείχατε σήμερα στην ε, συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ για τις λεπτομερεί απαντήσεις που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα. Όντως υπάρχει πολύ πεδίο δράσης ακόμα για, τον, για τους Ρωμά. Είναι ένα πρόβλημα πολύ περίπλοκο, το οποίο δεν έχει λυθεί ούτε σε εθνικό ούτε σε κοινοτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όλοι παρακολουθούμε ε, παρακολουθούσαμε την κρίση το καλοκαίρι του 2010 στην Γαλλία με τους ε, Ρωμά από τη Ρουμανία. Αυτό συζητήθηκε στο, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο εδώ και σε επαφές που είχαμε με τη γαλλική κυβέρνηση. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Πώς σχολιάζετε τις διάφορες ε, προσπάθειες κάποιων κρατών μελών να βασίζουν ε, την λύση της ένταξης στην, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ε, Σέγγεν με το θέμα των ε, Ρωμά. Ε, Σέγγεν λοιπόν και Ρωμά. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν μιλούμε για τους Ρωμά, μιλούμε για ένα λαό που έχει ή θα έπρεπε να έχει λάβει, να έχει υποστεί αρκετά καλά. Οι περισσότεροι όμως όταν μιλάμε για αυτούς μιλούμε για διακριτική μεταχείριση, μιλούμε για πράξεις ε, ε, βίας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν δράσεις ε, για να τους συμπεριλάβουν, να τους εντάξουν στην κοινωνία τους και να αποφύγουν τέτοια, τέτοιες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Η... Δεν υπάρχει... Οι Ρωμά λοιπόν δεν μπόρεσαν ούτε να επιλέξουν ούτε να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη. Μήπως όμως αυτό είναι λίγο μια προσπάθεια χειραγώγησης γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα που τους, αφορούν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Αν μπορέσετε να απαντήσετε και σε 10 λεπτά, θα μπορέσουμε έτσι και να ολοκληρώσουμε και την ημερήσια διάταξη που έχουμε για σήμερα. Ευχαριστώ. Αύριο θα είναι εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οπότε οτιδήποτε διοικητικό θέμα ή ερώτημα μπορείτε να το θέσετε σε αυτόν. Αυτό το θέμα δεν είναι άμεσης αρμοδιότητας του δικού μου Υπουργείου. Η μονάδα που είναι υπεύθυνη για τους ε, εθνικούς πόρους είναι υπεύθυνη για τέτοια θέματα. Αλλά το θέμα της κυρίας ε, Γκόνς ε, προφανώς είναι θεμητό, αλλά το θέμα της ε, κατακαιρματισμένη εκπαίδευση είναι θέμα Υπουργείου Παιδεία, όπω καταλαβαίνετε ε, και το πώ εντάσσονται τα παιδιά των Ρωμά στα σχολεία και πώ εκπαιδεύονται. Ε, βλέ, παρακολουθούμε και εμεί τα θέματα αυτά, αλλά το φάκελο αυτό, η οδηγία και τα υπόλοιπα θέματα που άπτονται αυτή ε, ανήκουν σε άλλα Υπουργεία και δεν είναι στη δική μου ορμοδιότητα Οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Τώρα, για την ένταξη. Κυρία Μπόσκουρτ, μου είπατε κάποια καλά λόγια όταν είπατε ότι ναι, προσπαθούμε να είμαστε ρεαλιστέ. Όντω, είναι σημαντικό να είμαστε ρεαλιστέ. όχι μόνο από τούτη τη σκοπιά. Αλλά και επειδή βλέπετε ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες κατά από τις οποίες ζουν οι Ρωμά στην Ισπανία, την Ιταλία, την ε, ε, Ρουμανία, την Ουγγαρία. Ε, υπάρχουν λοιπόν, διέπονται οι συνθήκε αυτές και από το τι συμβαίνει στην κάθε μια τοπική κοινωνία. Ε, τώρα, η ένταξη δεν μπορεί να γίνει και οι ξεχωριστές ας πούμε κατοικίες για τους Ρωμά σε συγκεκριμένες περιφέρειες δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το, μπορεί να το επιλέξει ένα κράτος μέλος θα έχει σίγουρα, δεν μπορούμε να το δούμε σαν κάτι ουδέτερο, δηλαδή αν αποκλείσουμε σε μία πλευρά της πόλης τους Ρωμά, αυτό θα έχει επιπτώσει. Ε, κανένας από τους Ρωμά δεν μπορεί να πάει σε ένα ε, ε, ειδικό σχολείο επειδή είναι Ρωμά ή επειδή είναι φτωχός. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η εξή. Υπάρχουν κοινότητες που περιμένουμε να συμβάνουν στην όλη προσπάθεια ένταξης. Ε, πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις κοινότητε, πρέπει να βοηθήσουν στην προετοιμασία όλων αυτών των δομών και πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες διαδικασίες διαχωρισμού. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις τοπικές κοινωνίες να αναλάβουν όλο το άχθος. Ε, υπάρχει, μιλούμε και, δεν μιλάω για χωριστή ε, εκπαίδευση, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτό να βοηθήσει τους φοιτητές, τους μαθητές, σε σχέση με την ένταξή του σε ένα φυσιολογικό σύστημα. Ε, στην ε, Ουγγαρία έχουμε το σχολείο Γκάντι που είναι ένα από τα ε, βασικά επιτυχημένα προγράμματα για τους Ρωμά. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες βεβαίως που θα υποστηρίξουμε. Ένα ειδικό είδος ας πούμε ε, εκπαίδευση ίσως να ήταν καλό για να υποστηρίξουμε τους μαθητές Ρωμά, να δημιουργήσουμε ίσως ε, ε, hostel για, τους, για τα παιδιά των Ρωμά για να μπορέσουν να μένουν, για να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, να πηγαίνουν στο ίδιο πανεπιστήμιο που πηγαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα για το σύστημα το φορολογικό, το flat rate. Αυτό είναι θέμα κρατών μελών. Βέβαια, ε, δεν μπορώ να τα πω όλα σε μία φράση, αλλά πρέπει να γίνουν όντω κάποια βήματα και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή η εισαγωγή ενός φορολογικού συστήματος ε, flat rate ε, είναι ένα από αυτά τα βήματα. Βεβαίως ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μα τι οικογένειε που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Τώρα, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν γίνεται ε, να, μην, να μην τρώει ας πούμε, ένα ζεστό φαγητό ένας, ένα παιδί το οποίο είναι φτωχό ή επειδή είναι Ρωμά. Ε, στα σχολεία, στο δημοτικό, τα παιδιά τρώνε ε, το μεσημέρι στο σχολείο. Ανεξαρτήτως του που ανήκουν και αν είναι καλοί μαθητές ή όχι. Άλλα σχολεία θα μπορούσαν ίσως να παρέχουν και ε, γεύμα το βραδινό. Μπορεί να σα ακούγονται λίγο αστεία αυτά που λέω, αλλά δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα στην ε, Ουγγαρία και το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να απαντήσω τώρα στην κυρία Κιγιόμ. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό όταν μιλούμε για το ευρωπαϊκή ε, στρατηγική πλαίσιο για τους Ρωμά. Υπάρχουν κρατημέλη όπου ζουν παραδοσιακά τα, κοινότητα στο των Ρωμά και υπάρχουν και οι χώρες στόχοι που θα ήθελαν είτε να πάνε οι Ρωμά είτε στέλνονται οι Ρωμά ε, εντάξει υπάρχουν πολλοί διάφοροι τρόποι να το πούμε αυτό αλλά ξέρουμε ότι η ελεύθερη κινητικότητα των πολιτών είναι μία από τι βασικές επιτυχίες της Ευρώπης και αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να επωφελείται. Κάθε πολίτης μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να μετακινηθεί και για οικονομικούς και για άλλους λόγους σε οποιοδήποτε μέρος της Ένωσης θέλει. Κανείς όμως δεν θα πρέπει να καταχράτε αυτής της ευκαιρίας για εγκληματικούς λόγους, για παράδειγμα. Αυτό δεν μπορεί να δίνει ευκαιρία σε κάποιους ε, λαθρέμπορους ε, είτε εμπόρους ε, ανθρώπων. Να διατηρήσουμε λοιπόν την μεγάλη αυτή επιτυχία της Ευρώπης, την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αλλά να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τι εγκληματικέ αυτέ συμμορίε, οι οποίες μεταφέρουν ανθρώπου από το ένα κρατο μέλος στο άλλο για να καταχραστούν των κοινωνικών συστημάτων των κρατών μέλων αυτών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν, αυτές τι δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματος θα πρέπει να τι έχουμε πάντα υπόψη μα. Πάμε πάλι πίσω στην οδηγία για, την, για, τις, για, τις διακριτικές, για τη διακριτική μεταχείριση. Αυτή η οδηγία είναι που θα μα βοηθήσει να πάρουμε περισσότερα μέτρα. Τώρα, η ένταξη της κοινωνίας των Ρωμά στην κοινωνία των υπολείπων. Το είπε νομίζω ο κύριος Μπρόγκς. Ε, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν υποκείμενα, όχι αντικείμενα όπως είναι τώρα. Πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο, πρέπει να είναι εταίροι μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε απτές αλλαγές. Και πρέπει να ενισχύσουμε τις οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Ρωμά. Οργανώνουμε δύο ε, ε, events στην, ε, στην ε, στην, στις Βρυξέλλες ένα το Φλεβάρι και ένα στην Ουγγαρία. δύο εκδηλώσεις. έτσι ώστε να έρθουμε κοντά με, την, με τις κοινωνίες των Ρωμά. η εκδήλωση αυτή θα γίνει στη Βουδαπέστη και θέλουμε αυτό, αυτή η εκδήλωση να μην είναι απλώς επαγγελματικό γεγονός. Θα είναι όμως η πρώτη φορά που θα μπορούμε να συζητήσουμε ε, πάνω στην ανακοίνωση της Κομισιόν γιατί θα διηγεί για τους Ρωμά. Θα είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Επόμενο ερώτημα τώρα. Βεβαίως είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει και μιλούμε για τις ε, χώρες που φιλοξενούν τους ε, ε, Ρωμά και τις χώρες προέλευσης των Ρωμά. Η διακίνηση, η ελεύθερη διακίνηση ναι είναι καλή, αλλά τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν εκεί όπου δημιουργούνται. Αυτές λοιπόν οι χώρες ε, έχουν σημαντική, σημαντικό ρόλο να παίξουν. Τα υπόλοιπα βεβαίως κρατημέλη δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους και να αγνοήσουν το πρόβλημα και ο Υπουργό που μίλησε πιο πριν αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, υπάρχει μια παρεξήγηση στη Δυτική Ευρώπη για τους Ρωμά. Θεωρούν ότι η κοινότητα των Ρωμά ε, ζει νομαδικά. Δεν είναι σωστό αυτό. Στη Ρουμανία, στην Σλοβακία, στην Ουγγαρία οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, σπίτια. Ε, μπορούν να θέλουν να μετακινηθούν από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά αν δεν θέλουμε να δούμε απλώ έτσι μεγάλους όγκους ανθρώπων να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε τη συμβολή και άλλων κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί από όπου δεν υπάρχουν, και όπου δεν υπάρχουν μεγάλες ομάδες Ρωμά για να βοηθήσουν τις ε, χώρε που έχουν σημαντικό πληθυσμό Ρώμα. Τώρα, πολύ σημαντικό επίσης ε, ερώτημα. Ε, πάντα πρόβλημα είναι τα χρήματα. Προφανώς τα κονδύλια δεν επαρκούν για να επιτύχουμε ποιοτική βελτίωση. Αλλά η νέα φάση της ε, χρηματοδότησης, ε, της οργάνωσης, ε, του σχεδιασμού χρηματοδότησης θα, πρέπει, θα ξεκινήσει τόσο λίγο. Οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους παλαιούς πόρους που έχουν διατεθεί, αλλά και με το κατά πόσο υπάρχουν νέοι. Πρέπει να δούμε κατά πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι πόροι και τι έγινε με τους πόρους τελικά που ήταν διαθέσιμοι. Χρησιμοποιήθηκαν για καλό σκοπό λήφθησαν από αυτούς που έπρεπε ή όχι. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολύ λεπτομερής αξιολόγηση επιπτώσεων και ανάλυση και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για μελλοντικού προϋπολογισμούς ή για διάθεση μελλοντικών πόρων ώστε να βελτιώσουμε δραματικά την ε, ζωή των Ρωμά. Και τώρα μιλώ εδώ και επενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, το Περιφερειακό Ταμείο δίνει κονδύλια για τη βελτίωση των ε, βιωτικών, του βιωτικού επίπεδου ε, των ανθρώπων αυτών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίω είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ξέρει κανεί αν τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ε, κονδύλια που του δίδονται. Οπότε τώρα θα δούμε κατά πόσο όλα αυτά από θεωρία γίνονται πράξη. Τώρα στην κυρία Ενετφέλτ, δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάτε, αλλά στα πλαίσια της ε, κοινωνικής ε, ένταξης είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ε, διακριτικής μεταχείρισης επί τη βάση της εθνικότητας, είτε στο χώρο εργασίας, είτε στις αρχές, είτε στο σχολείο. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους αξιωματούχους που χρειαζόμαστε και που έχουν να κάνουν με τους Ρωμά στην καθημερινή τους εργασία. Και επίση χρειαζόμαστε υποστήριξη. Χρειάζονται οι Ρωμά συγκεκριμένου ανθρώπου που να μπορούν να ε, εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά του καλύτερα όταν ε, έχουν, ένα, όταν έχουν έρθει σε επαφή με εθνικέ αρχέ. Τώρα για τη Σέγγεν. Θα να πω το εξή. Η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι αυτά τα δύο θέματα δεν θα πρέπει να συνδέονται. Η Σέγγεν και η ένταξη των Ρωμά δεν θα πρέπει να συνδέονται. Να συνδέονται. Είναι αντικρώμενε οι απόψει των κρατών μελών προ αυτό, αλλά εμεί είμαστε διατεθειμένοι να, να αγωνιστούμε. Ε, θα θέλαμε η, Ουγγαρ... η Ρουμανία συγγνώμη, και η Βουλγαρία να μπουν στην ε, ζώνη Σέγγεν. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολύ υψηλέ ελπίδε. Θα δούμε κατά πόσο ε, θα μπορέσουμε στου υπόλοιπου 6 μήνε να κάνουμε κάτι, αλλά Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνδέουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Κάποια κρατημέλη το κάνουν και αυτό είναι άσχημο. Ευχαριστώ. Θέλετε να αναφερθείτε και σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Χαίρομαι για τα ερωτήματά σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και εάν νομίζετε ότι θα ήταν χρήσιμο, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε στο τέλος της Προεδρίας. Μπορώ να παρευρεθώ εδώ και να σας προσκαλέσω σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ουγγαρία. Να σας δώσω τις πληροφορίες και ελπίζω να έχετε μια θετική εικόνα για την Ουγγαρία όταν ε, έρθετε στη χώρα μας. Βεβαίως κύριε Υπουργέ, συμφωνούμε όλοι και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούμε στενά με την ε, εκπεριτροπής Προεδρία, με την Ουγγρική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, είναι θέμα που μας απασχολεί, μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας. Η κοινωνική ένταξη είναι ένα στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και η καταπολέμηση βεβαίως των διακρίσεων. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν μιλάμε για τους Ρωμά στην Ευρώπη. Έχουμε μία συνεχιζόμενη συζήτηση και με μεγάλη μας χαρά να σας ακούσουμε στην Επιτροπή μας για τις εξελίξεις υπό την Προεδρία σας, να δούμε πώς ε, εξελίσσεται το όλο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για το χρόνο που διαθέσατε στην ε, Επιτροπή μας. Μας ε, σκιαγραφίσατε τις προτεραιότητές σας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους βουλευτές γιατί περιορίστηκαν στο χρόνο που έπρεπε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστούμε και πάλι.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα σημείο ακόμα και θα έχουμε χρόνο να το εξετάσουμε λοιπόν αφού είναι ένα σημείο. Σχετίζεται με την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ε, κύριες ε, προκλήσεις ε, με τα βασικά επιτεύγματα. Έχουμε αυτό το σημείο ακριβώς σήμερα που ακούσαμε για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε χθες στη Μόσχα. Καταδικάσαμε αυτή την τρομοκρατική επίθεση και βέβαια πρέπει να βελτιώσουμε τις κοινέ μας προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κοινοτικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής και πολιτικής. Θα έχουμε λοιπόν τώρα μια ανταλλαγή απόψεων πάνω στο έγγραφο εργασίας στην ανακοίνωση της Εκομισιόν σχετικά με την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για την αντιτρομοκρατική διαδικασία στρατηγική και πολιτική. Η συνάδελφο κυρία Σοφία Εντφέλντ έχει προετοιμάσει την εισήγηση αυτή. Θα μας κάνει μια παρουσίαση και μετά θα ανοίξει η συζήτηση ούτω ώστε τα άλλα μέλη να συζητήσουν το θέμα. Και ίσω μπορούμε να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν και την Προεδρία. Κάποιο σήκωσε το χέρι του από τη κυρία Σίμπιλ θέλει κάτι να παρατηρήσει διαδικαστικό. Go ahead. No, no, no. you were asking for the Α, ζητήσατε το λόγο. Α, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Εντιφέλ. Yes, thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στα χθεσινά γεγονότα και νομίζω ότι κάθε τέτοια επίθεση καταδεικνύει την ανάγκη μιας πολιτικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας που θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Αυτός είναι και ο απότερος στόχος. Όμως κατά τα τελευταία δέκα χρόνια παρόμοιων πολιτικών δεν έχει γίνει καμία αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Το έγγραφο εργασίας που είναι πρόδρομος του τελικού εγγράφου αναφέρεται στα τελευταία δέκα χρόνια, όχι ότι πριν δεν υπήρχε τρομοκρατία η αντιμετώπιση της, αλλά από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 έχει αλλάξει η κατάσταση άρδιν και ακριβώς επειδή έχει εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται αποτίμηση, σαφής αποτίμηση είτε πρόκειται για υποδομές, εκπαιδευτική πολιτική, οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια εποχή οικονομικής κρίσης και λιτότητας θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές μας και πόσο στοιχίζουν. Δυστυχώς οι πολιτικές αντιμετώπισης τρομοκρατίας δεν υπόκεινται σε, αυτή τη, σε αυτό το δημοκρατικό έλεγχο. Γι' αυτό είναι πολύ θεμητή αυτή η συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε μία εις βάθος αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προβαίνει σε μια πρώτη αποτίμηση. Χαίρομαι που υπάρχει κάτι συγκεκριμένο επιτάπητος, αλλά βλέπω ότι είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, διότι ανακεφαλαιώνει ορισμένα μέτρα που έχουν ληφθεί χωρίς να δει τον αντίκτυπό τους ως προς την αυξημένη ασφάλεια. Γιατί λαμβάνουμε μέτρα για την ασφάλειά μας για να δούμε κατά πόσο είμαστε πιο ασφαλείς. Αυτό το ερώτημα δεν απαντάται από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλώς ασχολούμαστε με μία κατηγορία μέτρων. Μιλάμε για συλλογή στοιχείων, η οποία, η οποία πολλές φορές αποκλείεται. Γιατί, αυτή, γιατί εδώ υπάρχουν ελλείψεις. Στο έγγραφο εργασίας θα πρέπει να πω ότι για γραφειοκρατικούς λόγους έχει, ξεχωριστεί, έχει χωριστεί στα δύο, αλλά είναι ένα έγγραφο εργασίας. Προσπαθώ να ορίσω ένα πλαίσιο, ένα ερωτηματολόγιο για την πλήρη αποτίμηση των μέτρων κατά της τρομοκρατίας. Δεν δίνω, δεν φτάνω σε συμπεράσματα, απλώς υποβάλλω τα ερωτήματα. Θα ήθελα να κάνω μια βασική σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να τη δεχτείτε, να γίνει μια εις αποτίμηση από ένα ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων να ασχοληθούν με θέματα ασφάλειας, προϋπολογισμού πολιτικών ελευθεριών και ούτω καθεξής, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως δεν ενδιαφέρεται σε μία ενδελεχή αποτίμηση. Καταρχήν θα πρέπει να μας απασχολήσει η αποτελεσματικότητα. Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα διότι θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο. Υπάρχει ασφάλεια. Δεν πρόκειται για μαθηματικούς υπολογισμούς. Δεν μπορεί να γίνει ποσοστοποίηση, γιατί αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποδοτικότητα των μέτρων, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο θα χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα εις βάθος. Να μην μας απασχολήσει μόνο η πρόληψη, αλλά και η έρευνα και η δίωξη. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη βασική κατηγορία που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το κόστος. Όπως σας είπα, σε καιρούς ε, οικονομικής λιτότητας θα πρέπει να γίνεται δημοσιονομικός έλεγχος, αυστηρός έλεγχος για να ελέγχουμε και το τελευταίο λεπτό που δαπανούμε αυτό γίνεται στο τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, αλλά δεν γίνεται το ίδιο για τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές. Πόσο μας στοιχίζουν. Εγώ δεν κρίνω κατά πόσο είναι πολύ ή λίγο. Θα ήθελα να ξέρω όμως πόσο στοιχίζουν από πλευράς εθνικών προϋπολογισμών αλλά και κοινοτικού. Το τμήμα μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μελετά το ζήτημα και ελπίζω ότι σε δύο μήνες θα έχουμε περισσότερα αριθμητικά στοιχεία για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το τμήμα δημοσιονομικών στοιχείων δεν μπορεί να μας δώσει ποσά, δυστυχώς. Επίσης, θα θέλαμε να ξέρουμε ο ιδιωτικός τομέας τι ποσοστό αναλαμβάνει, διότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα ανατίθενται όλο ένα και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, ε, τελεκόμ, οι ιδιωτικές εταιρείες λοιπόν αναλαμβάνουν ένα μέρος του έργου αυτού και να και το οικονομικό και διοικητικό κόστος αυτών των μέτρων. Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε το ύψος τη συνεισφορά. Σε ένα τρίτο στοιχείο που είναι αυταπόδεικτο είναι οι επιπτώσεις της αντιτρομοκρατικής πολιτικής στις πολιτικές ελευθερίες, στο, στο κράτος δικαίου. Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς και το, θα το δείτε και στο έγγραφο. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η λογοδοσία, ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία, διότι η αντιτρομοκρατική δράση δεν αφορά την ε, ε, εφαρμογή του νόμου, αλλά αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες συμμετέχουν και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος ή να επιμείνουμε σε θέματα λογοδοσίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εμβριακή κατάσταση μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διακίνησης Πληροφοριών. Βεβαίως δεν υπάρχει, δεν δίνεται δημοσιότητα στο έργο τους. Ε, βλέπω ότι μερικοί συμφωνούν μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες πρέπει να υπόκεινται έλεγχο. Πρέπει να λογοδοτήσουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε την Επιτροπή ΣΤΙΚΑΜ στο δικό μας ε, Κοινοβούλιο. Μία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το αντίστοιχο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι αν υπάρχει μία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών, θα πρέπει να υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος και εποπτεία. Και αυτή είναι μία από τις συστάσεις μου. Τέλος, εάν έχουμε τα αποτελέσματα μίας εκτενούς μελέτης, θα πρέπει να είναι η βάση των μελλοντικών πολιτικών μας. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματική η αντιτρομοκρατική μας ε, πολιτική, δεν πρέπει να ζητάμε την επανάληψή της. Θα πρέπει να δούμε τι κάναμε μέχρι τώρα και να βασίσουμε αυτή την πολιτική, τη μελλοντική πολιτική στα συμπεράσματά μας. Είδαμε τι έγινε στην Τινησία, τα, τις τελευταίες εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει, θα ισχύσει ενδεχομένως στην Αλιαγερία, στην Ιεμένη. Υπάρχει ένας αναβροασμός. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ως προς τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, θα συντάξουμε μία έκθεση με βάση το δικό σας input Βάση της ε, τακτής διαδικασίας. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης θα γίνει μια κρόαση για να ακούσουμε Ευρωπαίους και μη εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας. Μπορεί να καλέσουμε και Αμερικανούς εμπειρογνώμονες. και θα υποβάλουμε τροπολογίες μετά την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω και τη δική σας συνεισφορά. First, let's, let's... Καταρχήν, ας ακούσουμε από τους βουλευτές που... Ο κύριος Διαθεντεμέρα καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι θα έπρεπε να παρευρίσκουμε και σε μια άλλη επιτροπή αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τόσο σημαντικό το θέμα που θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Οι εχθροί της δημοκρατίας είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τις ιδέες τους πέρα από έναν κυρίαρχο λαό, πέρα από το κράτος δικαίου. Οι τρομοκράτες ε, καταφέρονται κατά της ανθρώπινης ζωής, επιτίθενται κατά του μοντέλου ε, ζωής μας και κατά του κράτους δικαίου. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις ασφαλείας των κρατών μελών θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη δράση τους. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας χρειάζονται ορισμένα στοιχεία. Γνώσεις και πείρα, αντικειμενικότητα, ορίζοντας βλέψεων, και να αναγνωρίζουμε την προτεραιότητα των εθνικών παραγόντων και των κρατών. Επίσης θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στο, στο ειδικό παράγοντα και στη ιδεοντολογία την προστασία δηλαδή των θυμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον συντονισμό των πολιτικών πρόληψης και πολιτικών απάντησης. Ο συντονιστής της καταπολέμησης τρομοκρατίας, η Europol, η Eurojust, το Κέντρο Αντιμετώπισης Κινδύνων και τα αρμόδια ε, οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών μελών θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όλες οι αντιτρομοκρατικές δράσεις θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών, μέσα στα πλαίσια του χάρτη θεμελιωδών και οικουμενικών δικαιωμάτων. Θα συνεργαστώ με την Σοφή για να υποβάλω τροπολογίες για τη δημοκρατική λογοδοσία και δημοκρατική εποπτεία, που είναι πάγια πρακτική στα κράτη-μέλη και της εύχομαι κάθε επιτυχία στην εργασία. Της ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπορσελίνο. Η κυρία, με συγχωρείτε. Πολύ με ενδιαφέρει αυτό το θέμα γιατί μου έχει ανατεθεί ένα έγγραφο για τη στρατηγική και εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε ως προς την έρευνα και τις αρχές, τις βασικές αρχές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισης δηλαδή των συνθήκων ασφάλειας στην εσωτερική ένωμη τάξη. Οπωσδήποτε μας ε, έχει σοκάρει η χθεσινή τρομοκρατική ενέργεια και μπορώ να πω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στην τρομοκρατία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όπως το οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα ε, μιλήσαμε με τον Υπουργό και υπάρχει, είπαμε, αιτιώδη συνάφεια μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να το μελετήσουμε πολύ προσεκτικά, διότι πολύ συχνά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες υπάρχει αυτή η συνεργασία ή πολλές φορές μία τρομοκρατική πράξη δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του, της οργανωμένης τρομοκρατίας. Χρειάζεται λοιπόν να προωθηθεί μία κοινή εργασία ως προς αυτά τα δύο θέματα, διότι η ζωή, η ασφάλεια και το μέλλον καθώς και η γαλήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε όλα αυτά τα στοιχεία. Ελπίζω να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία για να συνεισφέρουμε και εμείς επί του θέματος αυτού. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Νετφέλτ για, το, για τις ερωτήσεις που έθεσε. Όντως χρειάζονται πολλές απαντήσεις. Καταρχάς, ποιο είναι το αποτέλεσμα εκτός Ευρώπης ό,τι αφορά την, ε, την, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σήμερα ε, όλα αυτά χρησιμοποιούνται από ακτιβιστές, είδαμε στην Κένια τι συμβαίνει, στην Ουγκάντα, συμβαίνει σε πολλές χώρε χώρες. Τέτοια μέτρα οδηγούν σε ε, λογοκρισία του τύπου, σε καταστατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, κάνει, που χρησιμοποιεί ο κάθε, ο κάθε ακτιβιστής για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται, πολύ, φαίνεται περίτρανα και μας δείχνει ποιο είναι ο, τρό, ο, ο, κίνδυνος που υπάρχει με αυτά τα μέτρα. Η κυρία Νεφέλτ θέλει να ερευνήσει όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ίσως θα πρέπει να δούμε την απόσταση κάποιων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμοκρατίας γιατί ε, παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε σκεφτεί 10 χρόνια πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσω να πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο την κατάσταση, να την ξαναδούμε και ίσως να είναι και χρονική στιγμή η ε, σωστή για να αποσύρουμε κάποιες, κάποια νομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν καλό να το κάνουμε. Καταρχάς, να ζητήσουμε από την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δει ποιες περιπτώσεις παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγραφεί από το 2001 και να μας δώσει μια εικόνα και επίσης στο follow-up των πτήσεων της CIA. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Αναφέρομαι στη σύσταση 7, τη δική σας. Τώρα, το ερώτημα είναι πάντα πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Χωρίς να θέλω να πω αν είναι λίγα ή πολλά, ε, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, αλλά εσείς λέτε στο έγγραφο εργασία σας πόσο, πόσο κόστησε στις ιδιωτικές εταιρείες, πόσο κόστησε στους φορολογούμενους. Είναι ερωτήματα αυτά που έχετε θέσει και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει ένα σημείωμα από τον συντονιστή αντιτρομοκρατικών ε, μέτρων από το 2010 που λέει ότι το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης είναι επίσης σχετικό και σημαντικό στα πλαίσια της αντιμετώπισης του, της τρομοκρατίας. Είναι πολύ απλό να λέμε ότι η διακριτική μεταχείριση και η περιθωριοποίηση οδηγεί τα άτομα στην ε, τρομοκρατία. Η διαδικασία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Παρ' όλα αυτά, η καλύτερη κοινωνική ένταξη θα μπορέσει να ενισχύσει την μείωση των ανθρώπων αυτών που τίνουν ίσως ε, να ε, στραφούν προς την τρομοκρατία. Και εδώ το καθήκον μας λέει είναι να εξετάσουμε μια πολιτική αντιτρομοκρατική υπό το φως της διακριτικής μεταχείρισης. Νομίζω ότι κυρία Ινετφέλτ αυτό θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Θα μπορούσατε να το συμπεριλάβετε και εσείς στο έγγραφο εργασία σας. Τέλος, το σημείο κλειδί είναι ότι 10 χρόνια μετά το, την 11η Σεπτεμβρίου να καταλάβουμε τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Γιατί εξακολουθούμε να, να συζητούμε περί της ηθικής του θέματος και δεν συζητούμε περί του νόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Χάγκης. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η κατεύθυνση είναι σαφής ε, αυτού του εγγράφου εργασία. και πολύ λογική. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι πραγματικά επιστημονική η προσέγγιση που έχετε επιλέξει και σας συγχαίρω γι' αυτό. Χάρηκα πολύ που είδα λοιπόν το κείμενό σα και έχω δύο ερωτήματα να σα θέσω. Εντάξει, έχω κι άλλα, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο θα θέσω μόνο δύο. Ε, υπάρχουν δύο προβλήματα τα οποία θα ήθελα να δείξω. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το εξή. Η συζήτηση για την αντιδρομοκρατία επικεντρώνεται ε, σε κάποια βασικά στοιχεία. Σε, με τα περισσότερα από αυτά τα βασικά στοιχεία συμφωνούμε. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία ακόμα συζητώνται. Και υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν την ε, ιδιωτικοποίηση και την ασφάλεια και κατά πόσο υπάρχει ε, ανισορροπία μεταξύ αυτών των δύο και κατά πόσο μπορούν να βρεθούν λύσεις για να επανέλθει η ισορροπία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Συζητούμε τα θέματα profiling και ε, εξόριξης δεδομένων. Ε, πολλοί και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, λένε ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για να μην μπούμε, όταν εξηλέγουμε δεδομένα, για να μην μπούμε σε προσωπικά δεδομένα. Αλλά κάποιοι θέλουν να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια. Ε, γιατί και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων του καθενό. Εγώ είμαι στη δεύτερη κατηγορία πρέπει να πω. Νομίζω ότι η ασφαλεία είναι πολύ σημαντική, είναι σημείο κλειδί. η διαφοροποίηση το, του προσώπου της τρομοκρατίας που παρατηρείται τελευταίως, δεν μπορώ να πω τώρα σε πολλές λεπτομέρειε, αλλά πρέπει να την έχουμε υπόψη. Αν δεν θέλουμε να κάνουμε προφίλ τρομοκρατών, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιστημονικοί στην προσέγγιση που θα επιλέξουμε και στους ορισμούς που θα δώσουμε, όπως ακριβώς το κάνατε και εσείς στο κείμενό σας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια, ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτών των δύο. Και πρέπει να αιτιολογήσουμε το διαχωρισμό αυτό χωρίς να θέλουμε να απαγορεύσουμε το ένα και να επιτρέψουμε το άλλο. Επίσης, αμοιβαιότητα. Περιμένουμε από τη ΣΥΠΑ να μας δώσουν δεδομένα. Οπότε πρέπει να έχουμε κι εμείς μια αρχή, ένα φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει αυτά ακριβώς τα δεδομένα. Κάποιοι λένε ότι η Citizen ίσως θα ήταν όντως η πιο σωστή, ο πιο σωστός φορέας ή η Eurojust ή η Europol για να αναλάβει αυτό το καθήκον. Και για το σύστημα PNR Είναι καλό που η νέα στρατηγική λέει ότι δεν χρειάζεται νέο, καινούργια ευρωπαϊκή... Ε, μάλλον ε, με εκπλήσει το γεγονό ότι λέει το κείμενο ότι δεν χρειάζεται νέο, ευρωπαϊκό PNR. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν φύγονται στο έγγραφο αυτό ως ανεξάρτητα ε, επιστημονικά θέματα που θα μπορούσαν να συζητήσουν οι προγνώμενες και όχι το κοινοβούλιο. Και εντάξει, σε ένα βαθμό αυτό είναι σωστό, αλλά υπάρχουν τέτοιοι ανεξάρτητοι προγνώμενες. Μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από πολιτικές ομάδες, αλλά δεν είναι ανεξάρτητοι από τις δικές τους αρχές και αξίες. Εγώ έχω διαβάσει αρκετέ ε, μελέτες πρόσφατα για την αντιτρομοκρατική ε, δραστηριότητα και υπάρχουν πολλές απόψει μεταξύ διαφόρων επιστημόνων, όπως και μεταξύ των κοινοβουλευτικών. Γιατί σε βασικά σημεία κάποιοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα προσωπικά, τα ατομικά δικαιώματα. Κάποιοι τείνουν να προστατεύσουν το, την πτυχή της ασφάλειας. Εγώ θα μελετήσω τις μελέτες που θα εκδοθούν και στο μέλλον, αλλά φοβούμαι ότι τα προβλήματα θα επαναλαμβάνονται κάθε φορά που θα υποβάλλεται τέτοια μελέτη. Δυστυχώς όμως λύση δεν πρόκειται να βρεθεί. Και ένα ακόμη σχόλιο που αποτελεί και τη βάση για τη δεύτερη ερώτησή μου. Ναι, η Citizen θα πρέπει να, είναι, να θεωρηθεί ως εξωτερικός φορέας και μετά θα πρέπει να έχουμε και εμεί δικό μας ανεξάρτητο αυτόνομο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και στην Ουγγαρία και στην δική σα χώρα υπάρχουν, υπάρχει επιτροπή στο κοινοβούλιο συγκεκριμένη που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αλλά υπάρχει πρόβλημα γιατί τα μέλη αυτές, αυτής της επιτροπής ε, υπόκειται σε εθνική διαπίστευση ασφάλειας. αν υπάρχει τέτοιος έλεγχος και δεν έχει να κάνει με κριτήρια διαπίστευσης, τότε οι αξιωματούχοι ε, των μυστικών υπηρεσιών δεν θα μας δώσουν τίποτα ουσιώδες για να λειτουργήσουμε. Αλλά αν δημιουργήσουμε εμείς ε, μέσα σε αυτή την επιτροπή μία διαδικασία διαπίστευσης, υπάρχει μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μπορεί να σκανάρει να περάσει από τη διαπίστευση αυτή τα μέλη που θα βρίσκονται σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ε, επιτροπή. Εγώ θα ε, μελετήσω ε, και ευχαρίστω περαιτέρω το κείμενό και ευχαρίστω να συνεργαστούμε για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό θέμα προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καμιά φορά δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει ένας στόχος της τρομοκρατίας. Αλλά ο ένας στόχος ε, είναι ίσως να αμφισβητήσουν ε, τις αξίες μας και τη δημοκρατία μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε αθέλητα προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ε, καταρχήν όχι μόνο την ενιακή αποτελεσματικότητα των μέτρων, αλλά γενικά όλα τα μέτρα, αλλά και τις επιπτώσεις στους πολίτες, ε, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε κατά πόσον τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται και που ίσως είναι λογικά έναντι στον ΕΙΠΑ, ιδίως για την ανταλλαγή των στοιχείων, χρειάζονται κατά τον ίδιο τρόπο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε στενή συνεργασία αστυνομία και δικαστικού τομέα. Και έτσι πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε τα ίδια μέτρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως με τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα θα ήθελα να κάνω και κάποια παρατήρηση εξ ονόματος της συναδέλφου Άννα Χέλτ. Η συνάδελφο Αναχίλτ είναι σκιώδη για την κοινωτική πολιτική κατάσταση της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να είναι παρούσα εδώ. Θα ήθελα όμω να παρουσιάσω κάποια θέματα εξ ονόματό τη. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ ότι το έγγραφο εργασίας είναι πάρα πολύ καλό και υποστηρίζει τα, ο σημαντικό αριθμό ε, πάρα πολύ σπουδαίων θεμάτων, ιδίως το θέμα των βασικών δικαιωμάτων και την ανάγκη για περισσότερες αναλύσεις της σχέσης κόστους ωφελίας των σημερινών μέτρων. Ταυτόχρονα έχει όμως κάποια ερωτηματικά και θα ήθελα περισσότερες αναλύσεις και συζητήσεις για τα εξή θέματα. Πρώτον, περισσότερη διευκρίνηση των μέτρων που πρέπει να ευθυνθούν στο κοινοτικό επίπεδο ή στο επίπεδο κρατών μελών όταν δηλώνεται ότι τα κράτη-μέλη είναι οι κύριοι παίκτες αυτής της πολιτικής. Βρία συστήματα στο κοινωνικό επίπεδο με χαμηλή διαφάνεια είναι πολύπλοκα, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Βέβαια θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε την αρχή της επικουρικότητας. όσον αφορά τι διαφορετικέ απόψει των κρατών μελών για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τι διαφορετικέ του εμπειρίε με την τρομοκρατία. Κατόπιν. Η Ενάλυση Κομισιόν όσον αφορά το λεγόμενο profiling των παικτών και το θέμα των κοινοτικών δικαιωμάτων για τα βασικά δικαιώματα. Τέλος, αναφέρει και ήδη η έννοια της ε, δημοσίας ιδιωτικής εταιρικής σχέσης, όπου όσον αφορά το θέμα του διαδικτύου που θίγει και η Κομισιόν και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αναλυθεί εις βάθος. Mr. Strasser. Thank Vorsitzender. ευχαριστώ Είναι πραγματικά σημαντικό το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εξετάσει το θέμα αυτό και αυτό δεν καταδεικνύεται από τα φρικτά γεγονότα της ε, χθες αλλά και από το όταν οι πολίτες μας ε, παρεμποδίζονται στην ελευθερία κίνησή τους και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ευρωπαϊκός συντονισμός το πρέπει να ξεπεράσει α, το σημερινά δεδομένα και γενικά συνεργασία της Ευρώπης με τους εταίρους που ενδιαφέρονται για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό που γίνεται εδώ και τώρα αυτή η συζήτηση γιατί εδώ και δέκα περίπου χρόνια έχει αλλάξει ριζικά ο κόσμος σε αυτό το θέμα και αυτό είναι να κάνουμε μία καταγραφή του πού βρισκόμαστε, προς τα πού θέλουμε να προχωρήσουμε και πόσο. Έτσι, εξ ονόματος του ΕΛΚ θέλω να προσφέρω στην εισηγήτρια την πλήρη μας συνεργασία. Ω κοιόδης εισηγητής εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω για τη συνεργασία μου αυτή και προσωπικά. Και όσον αφορά το έγγραφό σας αυτή τη στιγμή δεν μπορώ παρά το αποθετικό βάση των γραπτών πληροφοριών. Εμείς προτιθέμεθα απόλυτα να συνεργαστούμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε κοινά συμπεράσματα. Στο έγγραφο αναφέρονται ορισμένες γενικές ε, γραμμές που συμφωνεί με αυτό το ΕΡΚ, μια βασική ε, πολιτική και όχι μέτρα ad hoc, τι ανάγκη να υπάρχει αξιολόγηση, η να για το λεγόμενο ΜΕΠ, όπου βλέπω ότι εμείς ζητάμε εδώ μόνο αυτό που μας υποσχέθηκε η Επίτροπος. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής συμφωνούμε νομίζω δεν θα ήταν απόλυτα σύμφωνο με αυτό που θέλουμε. Η ασφάλεια βέβαια κοστίζει. Φυσικά κοστίζει. Όπως και η πολιτική ασύλου κοστίζει. Η πολιτική κατά των διακρίσεων κοστίζει. Αλλά τι χρειαζόμαστε. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν χρήματα για την ασφάλεια, θα πρέπει η χρήση τους να είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες και θα πρέπει να βρεις το σωστό συγχειρισμό με ένα περιορισμό της ελευθερίας των πολιτών. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα να δούμε την αποτελεσματικότητα του κανονισμού για τα υγρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν αυτόματες διακρίσεις κατά πολιτών λόγω κάποιων αυτοματοποιημένων δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το 89% των πολιτών θα εξεταστούν από εμά. Όχι, το 2-3% είναι εκείνοι που θα μας απασχολήσουν και οι άλλοι θα πρέπει κατά να εξαιρούνται από αυτά τα μέτρα. Η ανακοίνωση της Κομισιόν δεν αναφέρεται καθόλου στο ρόλο των μυστικών υπηρεσιών. Συμφωνώ βέβαια με τους σε αυτό είναι σε μεγάλο ποσοστό εθνικό θέμα. Αλλά ένα τέτοιο έγγραφο, μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία δεν μπορεί να έχει υπόθεση αν δεν εξετάσουν και το θέμα της συνεργασίας με τις ε, μυστικές υπηρεσίες, και η ανάπτυξη μιας σχετικής πρακτικής. Από τις εθνικές ε, υπηρεσίες ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, οι βέλτιστες πρακτικές, κατά πόσο μπορούμε πραγματικά μια τέτοια υπηρεσία να την εξετάσουμε αυτόν να αφήσουμε να εργάζεται μυστικά αφετέρου. Είναι δυνατόν. Η πολιτική άμυνας και η εξωτερική πολιτική αφορά το θέμα βέβαια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να συνεργαστούμε με την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, πώς είναι κατανομημένες οι ευθύνες, ποιος κάνει τι και αν σκεφτείτε την στρατηγική ΝΑΤΟ που υιοθετήθηκε στη Λισαβόνα και αναφέρει το, το θέμα της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ε, το θέμα της ε, πολιτικής προστασίας επίσης και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνει ποιος, πότε και σε τι μεγάλο ποσοστό. Γενικά έχετε υποβάλει μια πολύ ε, φιλόδοξη έκθεση, αναφέρεται σε διάφορες προθέσεις, αναλύσεις, μελέτες, ακροάσεις και άλλα αλλά για να υπάρξει ένα απτό αποτέλεσμα θα πρέπει να καθοριστεί κάποια προτεραιότητα. Να δούμε τι χρειαζόμαστε καταρχήν, τι χρειαζόμαστε μετά και ίσως στο τέλος. Για άλλη μια φορά εξ ο μάθος μας θα ήθελα να τονίσω την πλήρη συνεργασία και καθώς επίσης ε, την προσπάθεια να υπάρξει ένα κοινό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να διακόψουμε στις 12.30 ε, και στις 3 το απόγευμα θα έχουμε αρκετές ώρες μπροστά μας και αύριο το πρωί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ουγγρικής Προεδρίας θα συζητήσουμε συναφή θέματα να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να μην ζητούμε συγγνώμη από τους διαμηνείς συνέχεια γιατί περβαίνουμε το χρόνο μας. Και να μπορέσουμε να ακούσουμε και από την Προεδρία και από την Κομισιό να μας βοηθήσετε. Σας παρακαλώ πολύ με το χρόνο. Κύριος Βός. Ευχαριστώ. Και εγώ θα υποστηρίξω το ότι όντω χρειαζόμαστε μια αντιτρομοκρατική στρατηγική ευρωπαϊκή. Μιλούμε για τη διατήρηση τη ελευθερία μα και τη δημοκρατία μα. Χωρί ασφάλεια δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Επομένω, η στρατηγική αυτή είναι απαραίτητη. Ε, φυσικά υπάρχουν πολλέ πτυχέ που είναι σημαντικέ. Εγώ απλώ θα ήθελα να μιλήσω για τι νέε τεχνολογίε. Εν τω μεταξύ έχουμε και αυτό το cyber wall και ε, τα θέματα της χρηματοδότησης, της ε, τρομοκρατίας, το έγκλημα στο διαδίκτυο, ε, στοιχεία δηλαδή τα οποία περιλαμβάνονται στην όλη, στον όλο τομέα των νέων τεχνολογιών. Το θέμα του κόστους επίσης, νομίζω ότι αυτό που δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σήμερα, μάλλον θα μας κοστίσει επιστημονικά του αργότερα στο μέλλον, για να, είμαστε, για να δράσουμε προληπτικά και θα το πληρώσουμε δύο και τρεις φορές. Ένα ακόμη σχόλιο για αυτά που είπε η κυρία Σαρκεντίνη. Ένα μεγάλο τμήμα των όσων ε, είπε δεν νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω. Στρατηγική αντιτρομοκρατίας δεν ήταν αντιστρατηγική, ήταν μια πολιτική δήλωση αυτή που έγινε, οπότε μάλλον θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο ουσιώδη. Στο ποιο είναι δηλαδή το μέτρο που θα μπορέσει να ε, μας δώσει μία, να μας βοηθήσει στην στρατηγική, σε μια αποδοτική στρατηγική για την, αντι, για την τρομοκρατία, ε, για τις διοκτικές αρχές, ε, για το τι γίνεται με το θέμα της λογοδοσίας και την ευθύνη που έχουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Sí, <coughs> quería decir θα ήθελα να πω ότι η ασφάλεια είναι ύψης της ε, σημασίας ε, μέσα στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής δράσης. Ίσως όμως αποτελεί μια ουτοπία, δηλαδή απόλυτη ασφάλεια. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Θα ήθελα να σας θέσω ένα απλό παράδειγμα που ίσως να μην έχει άμεση σχέση αλλά άπτεται του θέματος ασφαλείας γενικότερα. Ο αδελφός μου, ο Αλμπέρτο, ο, ο οποίος ζούσε στη Σεβίλη και ήταν αντιδήμαρχος, ε, δολοφονήθηκε από την ΕΤΑ μαζί με τη γυναίκα του. Αυτό το θέμα το Ξέρετε ότι το συνδέουμε με, την, ε, με τη βασκική χώρα, αλλά η ΕΤΑ δρά σε όλα τα μέρη της Ισπανίας. Εγώ λίγες μέρες πριν τον ε, ρώτησα αν φοβόταν και μου είπε όχι, όχι, είμαι ο 800ος στη λίστα που έχει κάνει η ΕΤΑ, αλλά σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε αφήνοντας τρία ορφανά παιδιά, παρόλο που ήταν στο κάτω μέρος της λίστας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταστήσουμε τους πολίτες ασφαλείς παρά το γεγονός ότι ο αδελφός μου ήταν πολιτικός και τύχανε προστασίας, μερικής τουλάχιστον. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Σοφή που αναλαμβάνει αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και να μην φυσθούμε μέσον για να προστατεύουμε πάντα τους πολίτες, είτε είναι πολιτικοί είτε όχι. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση διότι τα θύματα της τρομοκρατίας δεν αντιμετωπίζονται σωστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τους προσδώσουμε τη σωστή τους θέση και γι' αυτό νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να λάβουμε υπόψη και την οπτική γωνία του θύματος. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τρομοκρατία εάν δεν λάβουμε υπόψη και το θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας, αλλά μέσα στα πλαίσια της ε, ζυγαριάς αυτής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση του θύματος. Αλλά όσοι δεν έχετε γνωρίσει αυτή τη μάστιγα δεν ξέρετε τι σημαίνει τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει να έχουμε προκαταλήψεις ως προς την τρομοκρατία. Εάν έχετε προκαταλήψεις, τότε δεν θα καταφέρετε τίποτα. Διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσω να σας υποστηρίξω. Ο κύριος Πρόντς. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ προσεκτικός ως προς τα αίτια της τρομοκρατίας, γιατί πολλές φορές αιτιολογούμε μια κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να ε, δικαιολογήσει τη μαζική θανάτωση ανθρώπων. Πολλές φορές οι ε, ε, διοκόμενοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο οι Ισλαμιστές γιατί μιλάμε για το Ιράκ και το Αφγανιστάν ως ε, μουσουλμανικές χώρες και θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα του Ιράν μελλοντικά. Πιστεύω ότι ως προς τη σύραξη της Μέσης Ανατολής δεν θα πρέπει να έχουμε μονομερή προσέγγιση, γιατί αυτό το θέμα δεν αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Θα πρέπει να παραμείνουμε εκτός αυτού του θέματος. Επίσης, θα πρέπει να ε, διώκουμε κάθε τρομοκράτη, είτε είναι Ιρλανδός, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε στην Ισπανία ε, είναι κάποιος που προέρχεται από τη βασκική χώρα. Τον ε, οποιονδήποτε δηλαδή οι, οι, οι διώκτες και οι διωκόμενοι θα πρέπει να, είναι, να λαμβάνουν υπόψη οποιοδήποτε προφίλ τρομοκράτη, είτε είναι και ο δάσκαλος της γωνίας, ο οποίος ε, βαρέθηκε να ασχολείται με τη δασκαλία και μετατρέπεται σε τρομοκράτη. Δηλαδή θα πρέπει να διώξουμε την ε, τρομοκρατία υπό όλες τις, τις μορφές. Κυρία Ρόιτοβα. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αυτή την διάρθρωση της έκθεσης της ε, συναδέλφου. Υπάρχουν, γίνονται ορισμένες συστάσεις στο τελικό μέρος της έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω την πρόληψη και να πω ότι κάτι που δεν αναφέρθηκε ήταν η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων. ότι η τρομοκρατία χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να φτάσει στους στόχους της. Και αυτό είναι θέμα δικής μας ευθύνης σε αυτή την Επιτροπή. Δηλαδή θα πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και συμφωνώ με όσα ελέγξαν επί του θέματος. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα της πειρατείας στον κυβερνοχώρο διότι κλέβουν στοιχεία, υποκλέπτουν στοιχεία. Η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις επίσης. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το έγγραφο είναι τα μέτρα που λαμβάνονται και κατά πόσο υπάρχει ένα πραγματικό κίνητρο. Δηλαδή έχουμε και το θέμα των υγρών στις χειραποσκευές. Δεν νομίζω ότι είναι μία αποτελεσματική στρατηγική και νομίζω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε αυτή την όχληση των επιβατών ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φάρμακα που μεταφέρουν. Εγώ είμαι γιατρός και ξέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που ταξιδεύουν διότι πολλές φορές δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους ε, επί του αεροσκάφους. Θα πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε και σε αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας θα πρέπει να αναθέσουμε αυτά τα θέματα και στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους, ε, και τους hackers της, ε, του κυβερνοχώρου, Λάντφορντ. Λυπάμαι γιατί δεν ήμουνα στο πρώτο μέρος της παρουσίασης γιατί έπρεπε να ασχοληθώ με ένα άλλο ε, θέμα που σχετιζόταν με τα βασανιστήρια. Εν πάση περιπτώσει, στη σύσταση 6, στη στάση 6 και 7, εκεί που γίνεται λόγος για δημοκρατική εποπτεία των αντιτρομοκρατικών ε, μέτρων και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Νομίζω ότι αυτή η εργασία θα πρέπει να συμβαδίζει με μια συνέχεια που θα δώσει η ΛΥΜΠΕ και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να δώσουμε συνέχεια στην δραστηριότητα των κρατών μελών σε σχέση με την έκθεσή μας που είχε καταρτιστεί τρία χρόνια πριν και είχαμε συνάντηση και με την Άμνηστη και με τον ε, Μάνφρεντ Νόβακ. Έτσι ώστε να συνδεστεί αυτή η εργασία με αυτή τη Σοφίντ και στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο επιτροπών σε σχέση με την παράδοση και τα βασανιστήρια. Ως προς τη συστάση 1 και 2, που υποστηρίζω είναι ότι κατά την αποτίμηση της στρατηγικής κατά της τρομοκρατίας έχει μεγάλη σημασία να επανέλθουμε στο, στην ποινική οπτική γωνία, δηλαδή στην ποινική δίωξη. Γιατί στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, κατά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι αυτή η αντιτρομοκρατική δράση ε, ανελήφθη εκτός ε, νομικής προστασίας, εκτός αυτού του πλαισίου και θα πρέπει να την εντάξουμε στα πλαίσια ποινικών διώξεων, διότι ότι αυτός είναι και ο απότερος στόχος, δηλαδή να διώκονται και να καταδικάζονται οι τρομοκράτες και όχι να εξαφανίζονται ή να τους ε, κρατούμε, να τους φυλακίζουμε ή να τους βασανίζουμε. Θα πρέπει να, ισχύσει, να έχει ισχύ ο νόμος μέσα στα πλαίσια των ποινικών διώξεων. Η κυρία Σαρτζεντίνη αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προς την αναθεώρηση των ε, αντιτρομοκρατικών μέτρων. Εδώ υπάρχουν ε, διάφορα επιμέρους ζητήματα και έχουν σημασία τα εντάλματα συλλήψεων. Δηλαδή όλα τα μέσα εντάσσονται στην ε, έρευνα και τη δίωξη ανάκριση και δίωξη και δεν απαγκιστρώνονται από την ε, οπτική των ε, ποινικών διώξεων. Ως προς το profiling, εδώ και δύο χρόνια είχα αναλάβει μία έκθεση για να ελέγξουμε την νομιμότητα αυτών των πράξεων. Τίποτα δεν έχει γίνει στο μεταξύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το profiling είναι αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό, διότι αναχαιτίζει τη συνεργασία με τις ε, αστυνομικές αρχές. Ε, η ευφυής εποπτεία όμως είναι σωστή, δηλαδή με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν. Υπάρχει λόγος, ο λόγος αυτού του φακελώματος όταν έχουμε υποψίες. Ως προς τις βομβιστικές ενέργειες του Λονδίνου, του 2007 θα πρέπει να δούμε τι γνώριζαν οι μυστικές υπηρεσίε πριν από τη βομβιστική ενέργεια. Δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίε ήξεραν πράγματα τα, ε, βάσει των οποίων θα έπρεπε να είχαν δράσει για να προλάβουν τις βομβιστικές ενέργειες. Γιατί όπως είπε και ένας συνάδελφος, θέλουμε οι μυστικές υπηρεσίες να μιλάν στις αστυνομικές αρχές, δηλαδή να υπάρχει συνεργασία μυστικών υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών. Ευχαριστώ. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο μου. Λοιπόν, θα, ακούσουμε τώρα την κυρία Μορβέη και παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Ε, újféleképpen ε, közelíti meg a Κοιτάξτε, ε, είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτή την ε, νέα προσέγγιση στην αντιτρομοκρατία. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή η αστυνομία, οι κυβερνήτες παρεμβαίνουν, ελέγχουν ε, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ή τι, δεν μπορούμε να πετύχουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον στόχο της ανεμοκρατακρίας. Υπάρχει εντύπωση ότι όσο πιο πολύ παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή θα υπάρχει καλύτερα αποτελέσματα για την αντιτρομοκρατία. Όχι. Η πιο πολύ δράση θα ήταν να αποσύρουμε τους ε, στρατιώτες μας από το Ιράκ και το Αφγανιστάν και το λέω αυτό στη χώρα μου. Ας αποσύρουν τους Ουγγρούς στρατιώτες. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί που βρίσκονται και δημιουργείται ένας τεράστιος κίνδυνος. Ο τεράστιος κίνδυνος είναι στην νομοθεσία και στην εφαρμογή του νόμου υπάρχει ένα φαινόμενο που ε, προωθεί τους φόβους για την τρομοκρατία και έτσι ορισμένες ομάδες ε, έρχονται σε επίθεση της ε, κατά την αντιπολιτευτή τους εκτός του ε, κράτους δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από ένα συμβουλευτικό σώμα ίσως ε, σαν ένα παράδειγμα της δικής σας έκθεσής σας και αυτό το συμβουλευτικό σώμα θα μπορούσε νομικά να αναλύει όλα τα μέσα που υιοθετούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα νόμο στην, στην Ουγγαρία που αναφέρει σε άτομα που ενδεχομένω έχουν σχέση με την δημοκρατία. Αυτοί μπορούν να κρατηθούν, να ελεγχθούν, να ανακριθούν. Αυτό είναι απαράδεκτο σε μια δημοκρατία η οποία πρέπει να διαπαιτεί από το κράτος δικαίου. Και θα χαιρόμουν γι' αυτό να υπάρχει και ένα ανεξάρτητο σώμα δικηγόρων που θα ελέγχει τις διαδικασίες που υπάρχουν στην καταπολέμηση κατά της τρομοκρατίας. Στην, στην Ουγγαρία, παραδείγματο, υπάρχει μια μεγάλη υπόθεση μόνο κατά της λεγόμενης ομάδας Χουνέο που σχετίζεται με οικονομική διαφθορά σε σχέση της σχετικής πολιτικής της οποίας ηγείται ο κύριος Γεωργή Πουτεχάζη που είναι ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, το είναι αντικείμενο μιας ε, δικαστικής ε, επίθεσης ε, για τρομοκρατία βρίσκεται κάτω από πάρα πολύ κακές προϋποθέσεις κράτησης στη φυλακή και γι' αυτό λέω θα ήταν καλό να υπάρχει ένα εξάρτητο σώμα δικηγόρων που θα ελέγχει την κατάσταση η ομάδα αυτή θα μπορούσε παραδείγματος να ελέγχει τι γίνεται στην Ουγγαρία ποιοι είναι οι όροι κράτησης τι κάνουν οι εθνικές αρχές και κατά πόσον τα άτομα αυτά έχουν πραγματικά μια δίκαιη δίκη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίφερ, εκπρόσωπος Κομισιόν, έχει κάτι να πει για μερικά λεπτά. Πρωτού ακούσουμε την κυρία Ιντφέλτ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να δώσουμε κι εμείς έτσι κάποιες πρώτες απαντήσεις σε όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούστηκαν. Γνωρίζουμε απόλυτα την ε, σημασία που έχει ο δημοκρατικός έλεγχος στον τομέα της αντιδημοκρατίας και στο πώς μπορούμε να εξορθολογήσουμε την ε, όλη αυτή η δικασία χρησιμοποιώντα ε, τεχνικέ ε, υποδομέ, χρησιμοποιώντα ε, εμπειρογνώμονε. Καταρχάς, η ανακοίνωση που έχει υποβάλει η Κομισιόν τον Ιούλιο πέρσι είναι μια πολιτική αξιολόγηση και το λέει ρητά. Είναι πολιτική αξιολόγηση, όχι τεχνικό κείμενο. αυτών που έχουν εφαρ αυτά που έχουν ε, γίνει από τη στρατηγική που έχει ε, εγκριθεί από το 2005 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Λέγεται λοιπόν σαφώς ότι αυτή η στρατηγική εξακολουθεί να ισχύει και επίσης αναγνώρισε ότι στην ε, ανακοίνωση του Νοέμβρη την επόμενη για τα επόμενα χρόνια αναφέρονται ποιε είναι οι συγκεκριμένε πτυχέ για την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, η οποία και, λέει ότι είναι συγκεκριμένα πολιτική απόφαση και για τα επόμενα χρόνια. Για την ε, τεχνική τώρα και για το πώς θα καταγραφούν όλα αυτά από την πολιτική ανακοίνωση του, επόμε... του προηγούμενου χρόνου θα το δούμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο τώρα να γίνει κάτι τέτοιο. Παρόλο που εσείς μπήκατε στο έγγραφο εργασία σας σε πολλές λεπτομέρειες, ε, βλέπουμε ότι οι προσδοκίες για μια τέτοια ε, έρευνα είναι πιο υψηλές από το ίδιο το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Ας πούμε, η αντιτρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο που αλλάζει συνέχεια. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν παλιά δεν εγγυώνται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα του μέλλοντος. Δεύτερον, η πολιτική ε, αντιμετώπιση τρομοκρατίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης απλώς συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές. Πώς μπορεί κανείς να συμβάλλει, να, να ενισχύσει τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορεί να, να σταθμίσει τις παραμέτρους και πώς μπορεί να συνδυάσει το ευρωπαϊκό επίπεδο και τις ε, πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Ε, τα πράγματα πάνε καλά γιατί δεν είχαμε κάποια μεγάλη ε, τρομοκρατική επίθεση ας πούμε. Και τέλος, ποιος είναι ο ορισμός. Τι σημαίνει τελικά μέτρα αντιτρομοκρατικά. Είναι πολύ λίγα αυστηρή ταινία τα μέτρα αυτά. Ίσως ε, να θέλουμε να έχουμε ένα, ε, μια πολυσχηδή αντιμετώπιση μέσα στην οποία θα υπάρχει και η αντιτρομοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κρίνουμε ε, και σε ό,τι αφορά το διοικητικό αυτός και το κόστος τι ακριβώς θα πρέπει να δοθεί στις πολιτικές αντιτρομοκρατίες και πού πρέπει να μπει το όριο της πολιτικής ευθύνης. Η Κομισιόν λοιπόν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν θεματικές προσεγγίσεις όπως η παράλληλη ε, ενημέρωση που ανακοινώσαμε τον Ιούλιο ε, να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ανταλλαγή πληροφοριών στι εσωτερικέ υποθέσει και στη δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια τεράστια εικόνα την οποία να μην μπορούμε να διαχειριστούμε. Α πούμε, σήμερα το, ε, το απόγευμα θα συζητήσουμε το θέμα των προπομπών. Ε, νομίζω ότι και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία ε, πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να, ε, να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα κάποια πράγματα είναι ανέφικτα. Ακούσαμε τον ε, Ούγκρο Υπουργό σήμερα και η, ε, Προεδρία δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο από αυτό. Προς το παρόν, όχι. Ωραία, οπότε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Νετφέλτ. Σίγουρα θα είναι δύσκολο, αλλά θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να απαντήσετε σε όσα ακούστηκαν. Σύντομα. Δεν θα συνοψίσω τη συζήτηση, γιατί περισσότεροι ήμασταν παρόντες. Δύο σχόλια. Και να πω και κάτι στην Κομισιόν. Είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς ξεκινήσαμε να συζητούμε την αξιολόγηση των πολιτικών αντιτρομοκρατίας και η συζήτηση στο παρελθόν και η συζήτηση σιγά σιγά πάει στο πώς βλέπουμε το μέλλον. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι τώρα συζητούμε μια αξιολόγηση, όχι έναν, το σχεδιασμό μιας νέας στρατηγικής. Αυτό μπορεί να είναι το ε, επόμενο βήμα, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επόμενο βήμα. Δεύτερον, όπως είπε η κυρία Χιμένεθ, αυτό δεν θα πρέπει να είναι, δεν θα πρέπει να είναι ιδεολογική συζήτηση. Δεν έχω τίποτα εναντίον της ιδεολογίας, αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια η συζήτηση γίνεται επί τη βάση υποθέσεων και μάλιστα πολύ περίεργων και ε, τραβηγμένων υποθέσεων πολλές φορές. Ο, το στόχος του εγχειρήματο αυτού για πρώτη φορά είναι να έχουμε γεγονότα, συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί γίνονται διάφορες δηλώσεις. Είπε και ο, ο Υπουργός Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό PNR γιατί τώρα είναι πιο ασφαλές να πετάει κανείς εκτός Ευρώπης παρά εντός Ευρώπης. Ε, εντάξει, αυτό είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Δηλαδή, πού το βασίζεται αυτό. Μπορεί να υπάρχουν οι αποδείξει, μπορεί εγώ να κάνω λάθο. Αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια καμία από τα αιτήμα, κανένα από τα αιτήματά μα δεν ικανοποιήθηκε για την, ε, για την υποβολή τέτοιων αποδείξεων. Ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε στην δήλωσή σα Κομισιόν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να καταδείξουμε την αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα αυτών των πολιτικών. Ε, και στην ίδια πρόταση λέτε η στρατηγική αντιτρομοκρατία εξακολουθεί να ισχύει, άρα θα συνεχίσουμε με την ίδια τρομοκρατία. Με βάση τι? Με βάση τι? ακούμε τέτοιες δηλώσεις ότι οι, πολιτικοί, πολιτικές είναι απαραίτητες κτλ. Ναι, μπορεί να είναι απαραίτητες και σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό είναι απαραίτητες, αλλά ας μας δείξετε και με αποδείξεις. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άλλος τομέας πολιτικής θα, οι νομοθέτε σε κανέναν άλλο τομέα πολιτική θα μπορούσαν να περάσουν απλώ λέγοντα να χρειαζόμαστε ένα νέο σιδηρόδρομο ή μια νέα, ε, μια νέα ε, γέφυρα. Ε, δεν μπορούμε να σα πούμε γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπιστευτείτε μα γιατί είμαστε κυβέρνηση. Ε, δεν γίνεται αυτό, δεν περνάει. Υπάρχει χρειάζεται ένα κατάλογο, υπάρχει κατάλογο με συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απάντηση. Αν δεν μπορούν να απαντηθούν από την, ε, από την Κομισιόν, τότε να μην υποβάλλετε προτάσει λέτε ότι στο κείμενο, το κείμενο είναι πολιτική αξιολόγηση των όσων έχουν επιτευχθεί. Ακριβώς αυτό δεν είναι. Εσείς λέτε τι έχει αποφασιστεί, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και δεν λέτε, δεν αξιολογείτε πώς εφαρμόστηκαν. Γιατί αυτό είναι θέμα που ούτε καν το θίγω στο δικό μου έγγραφο. Μας φορτώνετε με μέτρα τα οποία είναι εξευθελιστικά που δήθεν είναι απαραίτητα και πήγοντα και τα λοιπά και δεν έχετε καν αξιολογήσει τι έχουμε πετύχει. Σήμερα, επί τη βάση του δικού σας κειμένου, δεν ξέρουμε αν είμαστε πιο ασφαλείς από όσο ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Με αποδείξεις. Ε, δίκιο έχετε που λέτε ότι είναι δύσκολο να έχουμε συγκεκριμένες αντικειμενικές παραμέτρους. Πρέπει να προσπαθήσουμε όμως. Ε, ζούμε σε δημοκρατία. Όλη αυτή η συζήτηση μιλά για την, γίνεται για την ε, προστασία της δημοκρατίας και των ε, θεμελιωδών μας ελευθεριών. Αυτό συζητάμε. Αν δεν πιστεύουμε στη δημοκρατία πια, αν δεν πιστεύουμε στη δημοκρατικό έλεγχο, στην λογοδοσία, στη διαφάνεια, τότε εντάξει, ας πάμε σπίτι μας. Αν παίρνουμε μέτρα τα οποία έχουν σημαντικό κόστος, αν παίρνουμε μέτρα και θα είμαι λίγο κοινική εδώ, υπάρχουν άνθρωποι που υποφελούνται ε, από τα ε, μέτρα αυτά. Κάποιο ε, παίρνει λεφτά. Εγώ είμαι φιλελεύθερη, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να, να πληρώνεται κάποιο. Αλλά να ξέρουμε ποιανού λεφτά ξοδεύουμε και για ποιο λόγο. Ποιανού την ελευθερία περιορίζουμε και για ποιο λόγο. Αν η Κομισιόν δεν μπορεί να μα δώσει απάντηση για κανένα από αυτά, ε, τότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Τέλος, είναι δύσκολο, λέτε, να διαχωρίσουμε τι ε, αμυγό ε, τρομοκρατικές, αντιτρομοκρατικέ πολιτικέ. Ε, τα περισσότερα μέτρα έχουν δικαιολογηθεί με την γενική ομπρέλα αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και έχετε δημιουργήσει εξουσίε για δημόσιε αρχέ οι οποίε είναι τελείω άσχετε με την αντιτρομοκρατία. Υπάρχουν κάποια μέτρα, τα οποία έχω μελετήσει εγώ λίγο πιο προσεκτικά από άλλα, και που λένε ότι η χρησιμότητα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας περιορίζεται πάρα πολύ και τα μέτρα χρησιμοποιούνται κατά 95% για πράγματα που είναι άσχετα με την τρομοκρατία. Είναι αυτό ακριβώς, αυτές ακριβώς οι πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουμε, γιατί μιλούμε για τα δικαιώματα των πολιτών μας, μιλούμε για την ασφάλεια των πολιτών μας και μιλούμε για τα λεφτά των πολιτών μας. Και το χρωστάμε στους πολίτες μας να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε εγώ βασίζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο, μια που όλοι οι συνάδελφοι ήταν ιδιαίτερο συνεργάσιμοι, και να καταλήξει σε μια λεπτομερή εντελεχή αξιολόγηση των όσων έχουμε κάνει στον τομέα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. that was quite an statement. This is an ongoing debate, but we have much exceeded our time, so we thank the interpreters. We thank the interpreters and uh, we thank you all, the participants of this long morning discussion